Bene. Buon pomeriggio a tutti. <laughs> Quindi buon pomeriggio a tutti quanti. Se possiamo accomodarci. Καλησπέρα σε όλους. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Αν δεν έχετε αντίρρηση, Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να ξεκινήσω τις σημερινές μας εργασίες υπενθυμίζοντάς σας ότι πρόκειται για μία προσθήκη στις 7 Νοεμβρίου μια συνεδρίαση φέτος στις αρχές της χρονιάς ε, είχαμε κάνει δύο ενδιαφέρουσες ακροάσεις για το έγκλημα στο χώρο της πληροφορικής, στο χώρο των υπολογιστών, όπου η συγγήτρια έκανε, η Μόνικα Ολμάιερ έκανε πολύ ενδιαφέρουσες ε, προτάσεις. Επίσης, έγινε η ετήσια συνεδρίαση με τα εθνικά κοινοβούλια για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για την εσωτερική ασφάλεια. Επίσης, θα ήθελα από πλευράς Προεδρίας να δείξω ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον ε, στο σεμινάριο που έγινε για να δημιουργήσουμε ένα χώρο ε, συνομιλίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και μέσα αυτό το χώρο θα υπάρξει μια επικοδομητική αντιπαράθεση, θα υπάρξει ανταλλαγή καλών πρακτικών και θα μιλάμε για το ρόλο των εθνικών και του Ευρωπαίου νομοθέτη. Μία πρόσταση θα υποβληθεί από τους ε, συντονιστές ε, της ΛΥΜΠΕΣ, τους συντονιστές των Εθνικών Κοινοβουλίων, που χρησιμοποιούν ήδη μια πλατφόρμα συντονισμού. Θα ήθελα τώρα για αυτές τις εργασίες, για τις οποίες μιλήσαμε λίγο, να δώσω το λόγο στον κύριο Μπορσελίν, στην κυρία Μπορσελίνου. Ευχαριστώ. Αυτή η δεύτερη συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μου άρεσε που τα Εθνικά Κοινοβούλια ζήτησαν να καταστεί μόνιμο αυτό το ραντεβού, ούτω ώστε να είμαστε ανατακτά διαστήματα σε ραντεβού και να ετοιμαστούμε για, το ενδιάμεση, για την ε, ενδιάμεση ε, αναθεώρηση του προγράμματος της Στοκχόλμης που θα γίνει το 2012. Επίσης, από το 2013 θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας. Επίσης, η Κομισιόν θέλει να συνεργαστεί με, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο σχέδιο έκθεσης σημειώνω ότι στις 19 τρέχοντος θα υιοθετηθεί από την Κομισιόν μία ανακοίνωση για την ε, πρώτη χρονιά της εφαρμογής της εσωτερικής ασφάλειας. Οι σκιώδεις εισηγητές στην επόμενη σύνοδο του Στρασβουργού θα συνεδριάσουν μαζί μου και θα παρουσιάσω το, έκθεση, το σχέδιο έκθεσης πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Επίσης, η Κομισιόν θα μας παρουσιάσει και ένα άτυπο πλαίσιο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ε, ούτως ώστε να αξιολογήσουμε τις ε, πρωτοβουλίες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για την ε, στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Επίσης, προσωπικά αισθάνομαι ικανοποιημένη για το υψηλό επίπεδο συνεισφορών από τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που πήραν το λόγο κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και με τους οποίους θα είμαι σε επαφή για τη συνέχεια των εργασιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μπορσελίνο. Πάμε στο τρίτο σημείο της ημερησίας διάταξης που αφορά την πρόσβαση των μεταναστών. Θέλετε το λόγο. Κύριος Λέντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ήθελα να λάβω το λόγο για τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου προηγουμένω. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση και κάποιες ερωτήσεις. Σήμερα το πρωί έλαβε χώρα μια συνεδρίαση του προσωπικού και συμμετέσχαν και μέλη της γραμματείας της ομάδας μου. Ένας από τους συνεργάτες μου μου είπε ότι αυτή η συνεδρίαση δεν θα μπορούσε να γίνει, αλλά στην πραγματικότητα έγινε αυτή η συνεδρίαση. Περί τίνος επρόκειτο. Επρόκειτο για τις ακροάσεις και τις αντιπροσωπίες τα ταξίδια των αντιπροσωπείων για το 2012. Εμείς κάναμε ένα, μια συγκεκριμένη πρόταση για την Κύπρο. Αλλά δεν βλέπω πια αυτή την πρόταση στο κατάλογο. Έχουμε πάρει ηλεκτρονικά ταχυδρομεία από άλλες πολιτικές ομάδες που μας λένε ότι σήμερα ήταν επικοδομητική η συνεδρίαση αυτή. Αλλά κανείς δεν μας ενημέρωσε για όλα αυτά. Θα ήθελα να ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Από τη μια μεριά μας λένε ότι δεν έγινε αυτή η συνεδρίαση, μετά μας λένε τι έγινε. Γιατί δεν μας κάλεσε κανένας, γιατί μας λένε ότι δεν έγινε αυτή η συνεδρίαση, όταν στην πραγματικότητα έχει λάβει χώρα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα και αυτό συγκεκριμένο θέλω να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο έχω αναφέρει ήδη πριν από δύο εβδομάδε. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μία γεγραμμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να πάρουν <clears throat> εκθέσει. Ξέρετε ότι είχαμε οργανώσει μία συζήτηση για το θέμα αυτό στο παρελθόν και μου είχαν υποσχεθεί ότι θα υπάρξει ένα υπόμνημα το οποίο θα υποβληθεί θα διανεμηθεί σε όλους τους βουλευτές και αναφέρεται στο σύστημα μορίων, βαθμών δηλαδή, που εξασφαλίζει την ε, ε, κατανομή των εκθέσεων μεταξύ των εισηγητών. Πότε μπορούμε να έχουμε αυτή την ε, νότα. Για το πρώτο ερώτημα, για τη συνάντηση στην οποία αναφερθήκατε, οργανώθηκε όχι από τη Γραμματεία. Για τη δυνατότητα των βουλευτών και των, των ανεξαρτήτων ειδικά να, να συμμετάσχουν στο, στην ακρόαση, χθες το συζήτησαν οι συντονιστές, έχουν, το βάλαν ούτως ή άλλως στην ημερήσια διάταξη και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια απάντηση σήμερα. Πάμε στο σημείο 3 που αφορά τους μετανάστες που βρίσκονται σε αντικανονική κατάσταση, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας σε 10 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Η συνεδρίαση αφορά μια παρουσίαση της έκθεσης, πρόσφατης έκθεσης, από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έγινε μια ανάλυση του Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανία, Ελλάδας, Ουγγαρίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Πολωνίας και Ισπανίας. Ε, είναι τμήμα αυτή η έκθεση ενός ε, προγράμματος ευρύτερου του οργανισμού αυτού για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών που βρίσκονται σε αντικανονική κατάσταση στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία πρώτη έκθεση ε, δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο και αφορούσε την ε, κατάστασή τους ε, όταν εργάζονται σε οικιακές εργασίες. Τώρα, με αυτή την έκθεση θα έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και θα δημοσιευθεί μέχρι το 2000, μέχρι το τέλος του 2011. Φυσικά, Η κυρία Λουντοβίκα Μπάμφη είναι η υπεύθυνη. Θα παρουσιάσει αυτή την έκθεσή της και εν συνεχεία θα δώσει το λόγο στους βουλευτές για να κάνουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κυρία Μπάμφη. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Μέλη της Επιτροπής ε, Πολιτικών Δευτεριών, σα ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω την εισήγηση αυτή σήμερα. Είναι μια εισήγηση στην οποία θα προαγώ και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα βασικά αποτελέσματα μία εκθέσεως που αφορά την υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα που όπως ξέρετε ε, είναι ευρωπαϊκή, είναι μια υπηρεσία που έχει την εντολή να προσφέρει αρρωγή στα θεσμικά όργανα και στα κρατή-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου για τα δικαιώματα. Συγκεκριμένα. Πρώτη για μια έρευνα που είναι τμήμα μιας ευρυτέρα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα για τους σε αντικανονική κατάσταση βρισκομένους μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που θα ήθελα να συζητήσω μέσα σήμερα είναι τα βασικά αποτελέσματα όσον αφορά την προσβασιμότητα εις της υπηρεσίας υγείας. Έχουμε 10 χώρες με τις οποίες ασχολούμαστε και δεν μιλούμε μόνο για εκείνους οι οποίοι δικαιούνται προσβάσεως, αλλά για το πώς έχει η κατάσταση γενικά στην πράξη. Και όχι μόνο με τους νομίμως διαμένοντες, αλλά με όλους για τις σχέσεις με τις δημοσιαρχές κλπ. Και οι χώρες που κάνουμε τη σχέσεις είναι Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Σουηδία. Το πρώτο το οποίο θα σας τονίσω είναι το εξής. Στις 10 χώρες στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έχουν προσφέσματα, αλλά μόνο σε πέντε από αυτέ. οι προσφέρονται δωρεάν αυτέ οι πρώτε βοήθειες γιατί επίση έχουμε κάποιε χώρε όπου θα πρέπει οι έγκυε να πληρώσουν 2.600 ευρώ για να έχουν τον τοκετό να γεννήσουν οπότε έχουμε τέσσερι χώρε παρόλα αυτά όπου και πρόκειται για τι καλύτερε. Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο αλλά και Ισπανία όπου η προσβασιμότητα παρέχεται και πέραν των πρώτων βοηθειών που η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια παροχή και δωρεάν. Όμως, στις χώρες όπου πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας αυτό δεν γίνεται δωρεάν, είπαμε ότι εδώ πέρα έχουμε ένα πράγμα πάρα πολύ σημαντικό που μπορεί να οδηγήσει εις κίνδυνο για τη ζωή των νομίμως διαμένων μεταναστών διότι ψάχνουν εναλλακτικές ας πούμε χρησιμοποιούν το βιβλιάριο ή την κάρτα κάποιου γνωστού τους, το οποίο φυσικά αποτελεί κίνδυνο. Τώρα εκεί όπου υπάρχει, όπως είπαμε, πρόσβαση και πέραν των Ισπανία, Γαλλία, δηλαδή Ιταλία και Γαλλία πέραν των πρωτοβοηθειών και εκεί υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν ταχθεί. Σε ορισμένε περιπτώσεις δύσκολα πληρώνται αυτές οι προϋποθέσεις. Πρέπει δηλαδή κάποιο να αποδείξει ότι μένει μονίμως και νομίμως επί τρεις ή έξι μήνες τουλάχιστον σε όλη τη χώρα. Επίσης δεν διαπιστώσαμε ότι παρά του ότι μπορούν να έχουν υπηρεσίες υγείας πέρα των πρωτοβοηθειών σε αυτές τις χώρες υπάρχουν ε, ορισμένες υπηρεσίες όπως η the ε, existence in some countries of reporting duties, that is the practice. Η αποκατάσταση. Η αποκατάσταση είναι που καμιά φορά δεν παρέχεται, οπότε πολλές φορές είναι θέμα νομοθεσία, είναι θέμα διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί όσον αφορά την ε, γνωστοποίηση της ε, περίπτωσης στις ε, υπηρεσίες αλλοδαπών. Δηλαδή τι γίνεται. Όπου υπάρχει κάποια πρακτική γνωστοποίηση στις υπηρεσίες αλλοδαπών φοβούνται μήπως τους απελάσουν. Οπότε αυτοί οι μη διαμένοντες νόμιμες μετανάστες φοβούνται να προσφύγουν στις υπηρεσίες υγείας. Έχουμε τώρα δύο πάρα ευάλωτες βαράτες ομάδες. Πρώτα-πρώτα οι έγκυες, δεύτερον οι ανήλικοι. Αυτές οι ομάδες δικαιούνται σύμφωνα με το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ειδική προστασία. Οπότε θα έπρεπε και στι 10 αυτέ χώρε να είχαν ε, κάλυψη και για τι έγκυε. Διαπιστώσαμε ότι και στι 10 εν λόγω χώρε. μπορούν να δικαιούνται κάλυψη στον τοκετό και στις 10. Όμως σε τρεις χώρες πρέπει να πληρώσουν και αυτό βέβαια είναι πρόβλημα. Επίσης, για κάλυψη πριν και μετά τον τοκετό, μόνο σε τέσσερα κάτι μέλη του παρέχονται σχετικέ υπηρεσίε. Τώρα, όσον αφορά του ανηλίκου, μα έγραψε το ότι μόνο σε δύο από τι δέκα χώρε μέλη έχουμε αυτού του ανηλίκου που δεν διαμένουν νομίμω στη χώρα, οι οποίοι έχουν τα δύο δικαιώματα όπω και οι ε, οι πολίτες της χώρας. Όμως, στις υπόλοιπες χώρες δεν ισχύει αυτό. Συνόδευτοι ανήλικοι έχουν επίσης ε, πρόσβαση στις περισσότερες υπηρεσίες υγείας. Κάμε συντεύξεις με πολλούς επαγγελματίες του κλάδου της υγείας σε αυτές όλες τις χώρες και τι διαπιστώσαμε, ότι κατά αυτούς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θέματα ηθικής και διοντολογίας όπως ο όρκος του Ιπποκράτη έρχονται σε αντίφαση με την αντίληψη την γραφειοκρατική ή που θεσπίζεται από τον νόμο όσον αφορά αυτά, αυτά, αυτά, αυτά τα πρόσωπα. Γιατί ακριβώς αυτές οι αντιφάσεις αποτελούν αντικίνητρο για τον κόσμο. Μην προσφέρει τόσο καμία όμως το θέμα είναι βέβαια και σε ποιε περιπτώσει παρέχονται δωρεάν υπηρεσίε υγεία ή όχι. Σε κάποιε χώρε η διαδικασία επιστροφή των εξόδων είναι περίπλοκη. Οπότε και εδώ έχουμε πρόβλημα. Ιδίω για αυτού που δεν διαμένουν νομίμω. Οπότε, αυτά είναι κάποια από τα λεπτά τη έρευνα που κάναμε και η υπηρεσία που σα είπα των δικαιωμάτων. Πες μια εβδομάδα τα δημοσίευσε όλα αυτά. Και όποιος θέλει να λάβει ένα αντίγραφο μπορεί να βρει αντίγραφο στην έξοδο τη αίθουσας. Όμως η υπηρεσία των δικαιωμάτων και θεμελιών δικαιωμάτων επίσης προδιοποιεί τη σε κάποιες συμβουλέ, σε κάποιες προτάσεις για το μέλλον. Οπότε μη διαμένοντας νομίζω σε μια χώρα θα πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο πρόσβαση. Όσον αφορά την αναγκαία περιθάλψη πέρα των πρωτοβοηθειών. Αυτό όμως δεν ακριβώ είναι πρώτη βοήθεια μόνο, αλλά θα πρέπει να καλύψει και άλλου είδου ιατρική βοήθεια, όπω α πούμε το να μπορούν να επισκεφθούν παθολόγο ή του γιατρού που χρειάζονται. Επίση, όσον αφορά τα ιατρικά έξοδα, και θα πρέπει να καλύπτονται και σε αυτό ακόμα και αυτού που δεν με νομίζω στη χώρα, ακριβώ όταν προβλέπεται και για του κατοίκου τη χώρα. Οπότε θα πρέπει να του επιτεύχονται τα έξοδα ή να υπάρξει ένα χωριστό ταμείο. Επίση, όσον αφορά τι προποθέσει όπω όπως την απόδειξη μόνιμη διαμονή για να μπορούν να πάνε στι όλα αυτά θα πρέπει να αναθεωρηθούν τόσο ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτέ οι προποθέσει δεν αποκλείουν τα πρόσωπα αυτά από τα δικαιώματά του ή στην ε, ιατρική πρόνοια. Τόσο αφορά την υποχρέωση κοινοποίηση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συλλέξουν τα δεδομένα από τι υπηρεσίε Ολοδαπών και δεν θα πρέπει να ε, υποχρεώσουν την, την, την, την ε, κοινοποίηση από μέρους των ιατρικών αρχών και των γιατρών και όλων των σχετικών με την ιατρική βοήθεια. Και τέλος, οι έγκες αλλά και οι ανήλικοι, αλλά και οι άλλες ευάλωτες ομάδες οι οποίοι δικαιούνται από όλα σε αυτών των δικαιωμάτων, θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. για τις πρωτοβάθμιες δευτεροβάθμιες ε, υπηρεσίες υγείας, ε, για το, για το υλικό που χρειάζονται όσον αφορά την κοίηση, αλλά επίση και, τα, και οι ανήλικοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να έχουν πρόσβαση, ακριβώς όπως και οι πολίτες της Χώρα. Αυτά θα ήθελα τώρα όμως, εν κατακλείδη, να σας πω τα εξή. Τον Μάρτιο του 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά έθεσε το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μη διαμενών των μεταναστών σε εκείνο το ψήφισμα όσον αφορά τα θέματα υγεία και τι ανισότητε. Και από την έγκληση στα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση ε, αυτών των προσώπων στι υπηρεσίε υγεία. Οπότε το δικαίωμα στη δημόσια υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Και αυτό καλύπτει και αυτέ τι ευάλωτε ομάδε. Διότι αυτοί δεν απολαύουν των ισών δικαιωμάτων, όπω οι άλλοι. Οπότε, παρακαλώ, λάβετε αυτό υπόψη στι ζυμώσει στο μέλλον. Και επομένω θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι στην προστασία αυτών των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά και περιμένω πώ και πώ τι ερωτήσει σα. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Λουντοβίγα Μπάμφη, λέει ο πρόεδρο, για όσα είπατε. Όσον αφορά την παρουσίαση αυτή τη έκθεση από την Υπηρεσία Θεμελών Δικαιωμάτων για αυτού του ε, μετανάστε που δεν διαμένουν μέσα στη χώρα ή σε αυτά τα 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο τον κύριο Γιακολίνο, ο οποίος και την καλοσύνη να αρχίσει την συνεδρίαση ή στην θέση μου. Εγώ ήμουν στο δρόμο από το αεροδρόμιο, διότι είχε καθυστέρηση το αεροπλάνο και συμπαθάτε μου. Τώρα, ήρθε η ώρα για τις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις προς την κυρία Μπάνθη όσον αφορά τα όσα μας είπε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα μεγάλο ενδιαφέρον την κυρία Μπάμφη. Θα ήθελα να κάνω κάποιες προτάσεις, αλλά και να μιλήσω για κάποιους προβληματισμούς. Εδώ εγώ δούλεψα στον ιατρικό κλάδο στην Ιταλία επί χρόνια. Και όλοι οι λαθρομετανάστες στην Ιταλία, τη στιγμή που μπαίνουν σε επαφή με την υγειονομική μας υπηρεσία, ε, τους δίνουμε ένα κωδικό. Αυτοί οι ξένοι που είναι προσωρινά στη χώρα μας, χάρη σε αυτόν τον κωδικό, μπορούν να εποφεληθούν από τις υγειονομικές μας υπηρεσίες, διαγνώσεις κτλ. Όμως ε, στην Ιταλία το σύστημα είναι πολύ περιοφυροποιημένο, όπως και πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο υγεία. Τελικά αυτές οι πληροφορίες τις έλαβε το Υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη ε, ότι η περίθαλψη ε, από περιφέρεια σε περιφέρεια στην Ιταλία διαφέρει. Αυτό που προκύπτει και αυτό που ξέρουμε είναι ότι το σύστημα συνολικά στην Ιταλία δεν είναι ομοιογενές. Υπάρχουν κάποιοι θύλακες αριστείας σε σχέση με την ε, γενική Ιταλική πραγματικότητα. Για αυτό το θέμα μια και εξετάσετε 10 κράτη-μέλη, θα μπορούσατε να δώσετε περισσότερε πληροφορίε, πιο λεπτομερείς πληροφορίε για την ε, κατάσταση του κάθε κράτου μέλου. Θα ακούσουμε όλε τι ερωτήσει και μετά θα απαντήσει η κυρία Μπάμφη. Κυρία Γκόνς, έχετε το λόγο. Πριν από κάποιου μήνε είχε λάβει χώρα μια συνδιάσκεψη για το ίδιο θέμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι απόψει των ΜΚΟ που έχουν μια ευρία εμπειρία για τα θέματα αυτά σε διάφορες χώρες και είχαν ουσιαστικά τα ίδια σχόλια, τα ίδια συμπεράσματα, τις ίδιες συστάσεις. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που βλέπω την έκθεσή σας και εφόσον καλύπτεται 10 κράτη-μέλη, ε, τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να είναι αντίστοιχη και η κατάσταση στα άλλα κράτη-μέλη. Ε, κατανοώ αυτό το οποίο λέτε ότι είναι κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο να, να προκύπτουν ανάγκες για περίθαλψη πριν από τον τοκετό και μετά από τον τοκετό στην περίπτωση των ατόμων αυτών που είναι σε μη κανονική κατάσταση. Θα πρέπει να καταλήξουμε κατά την άποψή μου σε ένα πακέτο το οποίο αποτελεί το ελάχιστο πρότυπο προστασίας και περίθαλψης και εφόσον είναι και η Κομισιόν εδώ θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη της Κομισιόν για το αν θα μπορούσε να υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα για την περίθαλψη που θα πρέπει να δίδεται σε όλου ανεξαιρέτω και πώ θα μπορούσε να επιληθεί το πρόβλημα χρηματοδότηση, αν χρειάζεται να υπάρχει ένα ειδικό ταμείο για να καλυφθεί αυτή η παροχή των υπηρεσιών και κατά πόσο μπορούμε να δώσουμε μια ενιαία λύση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. <coughs> Μούλτερ. Ευχαριστώ. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την παρουσίαση της κυρίας Μπάμφη. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Υπάρχει κάποια μορφή συσχετισμού μεταξύ των χωρών και του υγειονομικού επίπεδου περίθαλψης που παρέχουν και του αριθμού των μεταναστών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν υπάρχει υψηλό αριθμό παράνομων μεταναστών σε μια χώρα, αν αυτό έχει επίπτωση στην ποιότητα τη περίθαλψη. Οι χώρε που έχουν το χαμηλότερο αριθμό παράνομων μεταναστών είναι ίσω αυτέ οι οποίε έχουν καλύτερες παροχές και παρέχουν πιο εύκολα αυτές τις υπηρεσίες. Ένα δεύτερο στιγμίο. Εξεπλάγει που είπατε ότι σε πολλές χώρες δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη για περίθαλψη. Τι γίνεται για αυτούς που αρρωσταίνουν. Τους αφήνουν στην τύχη τους. Κύριος Κλής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την ορολογία παράνομος μετανάστης για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Δεν μιλάμε για χωρίς έγγραφα μετανάστες ή οτιδήποτε τέτοιο, μιλάμε για παράνομους. Ας τα λέμε τα πράγματα σίκα σίκα και σκάφη σκάφη. Με το όνομά τους. Στην Ευρώπη λοιπόν, κανείς κύριε Πρόεδρε <clears throat> δεν έχει αντίρρηση στο οι παράνομοι μετανάστες να έχουν πρόσβαση σε έκτακτες υγειονομικέ υπηρεσίε. Κανεί δεν το λέει αυτό το πράγμα ότι δεν πρέπει να γίνει. Αλλά θέτω το εξή ερώτημα. Ποια είναι η δική σα εντολή αυτή τη στιγμή. Κατά τη δική μου άποψη, η δική σα εντολή είναι να εξασφαλιστεί ο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ νομίζω ότι εσεί έχετε δώσει μια διασταλτική και για μένα απαράδεκτη ερμηνεία τη εντολή σα. Δίνετε συστάσεις και συμβουλές που έχουν σαν αποτέλεσμα τα νοσοκομεία τα οποία αντιμετωπίζουν παράνομους μετανάστες που θέλουν υγειονομική περίθαλψη να μην μπορούν να κοινοποιήσουν ε, το γεγονός αυτό στις αρμόδιες αρχές. Αυτό σημαίνει ότι εσείς παρεμβαίνετε σε αρμοδιότητες κρατών μελών και εμποδίζετε μερικά κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση. Γιατί είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς αυτό το φαινόμενο. Όταν κανείς απευθύνεται σε ένα υγειονομικό φορέα, είτε είναι δημόσιος είτε, δεν είναι, είτε ημιδημόσιος, είναι απόλυτα λογικό να πληροφορείται και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ισοτερικών. Δεν καταλαβαίνω γιατί εσείς προτείνετε να τροποποιηθεί αυτό. Όλα αυτά δημιουργούν την εντύπωση ότι το να <clears throat> πληροφορήσει κανείς τις αρχές για την κατάσταση αυτών των ατόμων είναι παραβίαση των δικαιωμάτων του, στο θεμελιωδών μα. Αν είναι παράνομη, είναι παράνομη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα και γι' αυτό πρέπει να είναι ενήμεροι. Αφού του δοθούν βέβαια οι απαραίτητε υγειονομικέ υπηρεσίε. Λοιπόν, δεν πρόκειται επομένω για καμία παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών να ανακοινώνεται αυτό, όπω δίνετε την εντύπωση εσεί. Κύριε Χέτ. Ευχαριστώ. Εγώ συγκλονίστηκα από αυτά που άκουσα. Τόσο που ξέχασα τι θέλω να πω. Εδώ μιλάμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υπερασπιστεί αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ καθυστέρησα όπως και εσείς ε, λόγω της καθυστέρησης του αεροπλάνου μου και δεν άκουσα όλη την παρουσίαση της κυρίας Μπάμφη. Αλλά συνειδητοποιώ ότι ο οργανισμός αυτός κάνει συστάσεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό το κατάλαβα. Εγώ φαντάστηκα ότι εδώ πρόκειται για μία έκθεση της, του οργανισμού και συνεχεία τα κράτη-μέλη θα κάνουν συστάσεις τα ίδια. Δεν νομίζω ότι είναι δουλειά του οργανισμού να κάνει συστάσεις. Έτσι. Ήθελα να το πω αυτό. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κατοχυρώσει αυτά τα δικαιώματα, όπως είπε η συνάδελφος προηγουμένως, αλλά επίσης ως δεδομένο ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών η παροχή τέτοιων υπηρεσιών, τι συστάσεις μπορεί ο οργανισμός σας να κάνει προς τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουν τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, τις οποίες εσείς βρίσκετε ότι δεν είναι ικανοποιητικέ. Και επίσης, αν έχετε εμπειρία από προηγούμενες μελέτες, αν έχετε προσέξει να βελτιώνεται αυτή η κατάσταση, αν η τάση είναι προς βελτίωση ή εν ώψη και των ροών των μεταναστών που έχουμε σήμερα, τα πράγματα χειροτερεύουν. Πρώτα πρώτα θεωρώ ότι στον τομέα της δημοσίας υγείας ε, έχουμε ε, προκειμένου έναν στενό ρυθμό σε σχέση με το τι εστί θεμελιώδη δικαίωμα, τι εστί συμφέρον της κοινότητας όσον αφορά το να υπεραμείνεται κανείς των δημιουργών δικαιωμάτων των μεταναστών ή από την άλλη μεριά τι νόμιμε θεμητέ προσδοκίε τη κοινωνία. Εν γέννη, διότι όταν μιλούμε για πρόσβαση ει το σύστημα υγεία, δεν εννοούμε μόνο τα δικαιώματα κάποιου φυσικού προσώπου μετανάστου. Μιλούμε γενικώ για την δημοσία υγεία. Επομένω, αν κάποιο δεν πάει στο νοσοκομείο και έχει μια πάρα πολύ μολυσματική μεταδοτική ασθενή αλλά δεν πάει στο νοσοκομείο διότι φοβάται ότι θα τον διώξουν ή ακόμα χειρότερα ότι θα τον δώσουν στις αρχές και μετά θα τον απελάσουν. Αυτό παραβιάζει τα δικαιώματα του μετανάστου. Αλλά όχι μόνο αυτό. Πρόκειται και πρόβλημα δημοσίας υγείας για όλους σε αυτή την κοινωνία. Επομένως, για πραγματικά μας ενδιαφέρει το συμφέρον της κοινωνίας θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο σκοπός του Συστήματος είναι να καλύψει ε, υπηρεσίες υγείας και επίσης να εξασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά ε, στάνταρ ε, υγειονομικής κάλυψης. Δηλαδή δεν είναι θέμα του τι θα κάνουμε με την ε, λαθρα, λαθρομετανάστευση, δεν είναι μόνο θέμα να διώξουμε του μετανάστε. το θέμα είναι το ότι θα πρέπει α πούμε μια επιδημία να ανασχεθεί και να μην εξαπλωθεί επομένω εμένα με συγκλονίζει, με, με, με σοκάρει το ότι έχουμε εδώ μια χώρα από τις αναλυθήσεις, στην Γερμανία εν όπου υπησχύει η πρακτική της γνωστοποίησης ή στις αρχές του καθεστώτος που διέπει κάποιον πάρει στο νοσοκομείο, κάποιον μετανάστου. Και ενδεχομένως αυτός απελαθεί. Η στη δική μου χώρα Προσπαθούμε, παλεύουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο να τους πείσουμε όταν είναι άρρωστοι να πάνε στο νοσοκομείο πέραν του αν είναι παράνομοι ή διαμένουν νομίμως. Οπότε έτσι λαμβάνουμε υπόψη και καλύπτουμε το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας. Πέραν των συμφερόντων και δικαιωμάτων του νόμιμου παρανομικού μετανάστη και τώρα. Θα έρθει η διαμενουν νομιμως οποτε ετσι λαμβανουμε υποψη και καλυπτουμε το γενικοτερο συμφερον της κοινωνιας περαν των συμφεροντων και δικαιωματων του νομιμου παρανομου μεταναστε και τωρα θα ερθει η ωρα να ψηφίσουμε σε λίγα λεπτά. Ε, έχουμε και την έκθεση τη αδέλφου Φλότρο, οπότε θα πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσο θα ακυρωθεί ή όχι η σύμβαση αυτή για τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών ε, του. Κάτι το οποίο κρεμεί πάρα πολύ καιρό. Οπότε θα πρέπει να, να κρεθεί το αν θα γίνει κύρωση τη συμβάσεω ή όχι. Οπότε, σα ερωτώ, τι θα γίνει με αυτό του είδου το, το FRA. Τι θα γίνει όσον αφορά την προσβασιμότητα στα στις υπηρεσίες υγείας. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος. Στην πολιτική. Χρησιμοποιούμε εφημισμού, όπω α πούμε λέμε, ε, ιδίω όταν λέμε για έλεγχο τη ελεύθερη σκέψη, όταν θέλουμε τον έλεγχο. Οπότε, πάρα πολλέ ε, αυτό το να λέμε το πέρα αντικανονική κατάσταση, αυτό είναι, είναι, είναι τερατώδες. Δεν θέλετε να πείτε παράνομη. Δεν το λέτε, δεν θέλετε. Αφού δεν θέλετε, τότε να πείτε κάτι άλλο το οποίο είναι ξεκάθαρο. Ξέρω εγώ, αυτή τον οποίο δεν έχει εγκριθεί η παραμονή, οπότε θα πρέπει να δούμε. Ε, Ποιο έχει βοηθήσει. Ε, αυτοί οι παράνομοι δεν έχουν εισφέρει τίποτα στο σύστημα και επομένω θα πρέπει να, να δούμε τι θα κάνουμε. Ε, η γενοδορία τι είναι. Η γενοδορία όταν κάποιο δίνει όταν βγάζει λεφτά από την τσέπη του και τα ξοδεύει για κάτι που αξίζει ή που δεν αξίζει. Εάν περισσεύουν κάποιοι πόροι, κάποια χρήματα, κάποιος επομένως θέλει να πρέπει να πάει στο γιατρό, φυσικά τότε ποιος να πει όχι, για όποιον και να πρόκειται. Αλλά συνήθως η ζήτηση είναι περισσότερη από όσο είναι προσφορά στον πρώτη υπηρεσία υγεία. Και έχουμε λίστες αναμονής για τις αυτές τις υπηρεσίες και στην Ηνωμένο Βασίλειο. Να είχαμε μια περίπτωση καρκίνου του δέρματος που θεωρείται πάρα πολύ ακριβό και επομένως όποιος δεν έχει εισφορές τότε δεν θα καλυφθεί ή δεν θα του κάνουν την αγωγή ή θα περιμένει. Θα ήταν πάρα πολύ γενναιοδρόντος να λέγαμε σε κάποιον ε, που έχει δώσει φορές να, να μην ε, περάσει από τη θεραπεία αλλά να πάει κάποιος πάνω όμως στους μετανάστες. Οπότε αυτό καταλήγει να μην είναι γενναιοδορία. Αυτό είναι προδοσία. Είναι κλοπή. Εγώ όμως σας προτείνω οι ευρωβουλευτές οι οποίοι είναι υπέρ του να καλυφθούν ιατρικά οι λαθρομετανάστες να φτιάξουν ένα ταμείο. Το ταμείο από το μισθό του και να καλύψουν το κόστο τη κάλυψη του λαθρομετανάστη. Αυτό θα ήταν κοινόδρο, αλλά δεν του βλέπω να το κάνουν. Ακούσατε κυρία Μπάνφη διάφορε ερωτήσει. Ορισμένε ερωτήσει. Έχουμε προβλέψει και μια ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα. Θα πρέπει να αρχίσει, να αρχίσει στις 4 ε, παρατέταρτο. Επομένω, κυρία Μπάμφη, θα ήθελα να σα δώσω 10 λεπτά ε, για να απαντήσετε σε όλε αυτέ τι ερωτήσει, για να μην καθυστερήσουμε την ε, ψηφοφορία. Σα ευχαριστώ για τι ενδιαφέρουσε ε, ερωτήσει. Να απαντήσω στον κύριο Γιακολίνο καταρχά. Ναι, κάλυψαμε σε κάποιο βαθμό και τι περιφερειακέ διαφορέ στο εσωτερικό μια χώρα. Η Ιταλία, α πούμε, είναι μία από τι χώρε που έχει τι μεγαλύτερε διαφορέ στο εσωτερικό τη σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη προς τους μετανάστες σε αντικανονική κατάσταση. Γιατί κάθε περιφέρεια τους αντιμετωπίζει διαφορετικά. Αλλά η έρευνα ε, έγινε σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Ήρθαμε σε επαφή δηλαδή με επαγγελματίε και με α, στη Λομβαρδία και στην Εμίλια Ρωμάνια. Ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ε, διάφορε από περιφέρεια σε περιφέρεια προ τα δικαιώματα και το καλύπτουμε στην έκθεση. Ε, ένα από τα βασικά θέματα είναι ότι η πρόσβαση στο γενικό παθολόγο δεν προβλέπεται σε όλες τις περιφέρειες, ενώ η πρόσβαση στο νοσοκομείο γενικά προβλέπεται σε όλες τις περιφέρειες. Σε ό,τι αφορά την προγεννητική και μεταγεννητική υπερίθαλψη, θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν κάποιες κοινέ διατάξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάποιες κοινέ προκλέψεις Θέλω να σας επενθυμίσω, όπως μας είπαν και εμάς, ότι εμείς ως οργανισμός δίνουμε στοιχεία. Εν συνεχεία, με βάση αυτά τα στοιχεία, υπάρχουν άλλα όργανα, άλλοι φορείς που είναι αρμόδιοι για να επεξεργαστούν αυτά τα στοιχεία για να καταρτήσουν ε, προτάσεις για πολιτική. Αλλά πιστεύουμε ότι οι έγκυες γυναίκες και οι μητέρες είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες ομάδες και πρέπει να προστατεύονται και αυτό που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι αυτή η προστασία δεν χορηγείται πάντα, άρα κάτι θα πρέπει να γίνει γι' αυτό. Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στον αριθμό των λαθομεταναστών σε μια χώρα και στο επίπεδο της περίθαλψης ε, που τους παρέχεται. δεν, από τα στοιχεία δεν προέκυψε κάποιο κάποιος συσχετισμός. Τώρα τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν ε, έκτακτη περίθαλψη. Αποκλείονται την επίγουσα περίθαλψη όταν δεν τους δίνεται. Αποκλείονται γενικά από το σύστημα υγείας. Καλό ερώτημα. Ε, το δικαίωμα στην επίγουσα περίθαλψη ε, ισοδυναμεί το δικαίωμα στη ζωή. Αν δεν έχουν ε, πρόσβαση σε αυτή την περίθαλψη δεν μπορούμε να φανταστούμε τι του συμβαίνει. Έγινε ένα σχόλιο ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε συστάσεις. Δεν κάνουμε συστάσεις. Δίνουμε συμβουλές με βάση τα στοιχεία που έχουμε και αφήνουμε τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν μόνα τους για το πώς θα εφαρμόσουν αυτές τις συμβουλές που τους δίνουμε μέσα στη δική τους εσωτερική πραγματικότητα. Φυσικά η έρευνα μεταφράζεται σε βήματα για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Ε, και πρέπει να ακολουθηθεί από κάποια βήματα. Συμφωνώ ότι η υγειονομική υπεριθαλψη είναι θέμα ολόκληρης της κοινότητας. Το να έχουν πρόσβαση οι μετανάστες στην υγειονομική υπεριθαλψη είναι θέμα που αφορά και την υγεία ολόκληρης της ε, κοινωνίας, ολόκληρης της κοινότητας. Τέλος, για την έλλειψη των πόρων, για αυτό το επιχείρημα που ακούσαμε, περί πόρων η παροχή περίθαλψης είναι και θέμα προϋπολογισμού, κονδυλίων, χρημάτων διαθέσιμων. Αλλά αν δίνουμε τέτοια περίθαλψη, ε, πέρα από την ε, κατεπίγουσα, θα μας βοηθήσει να ξοδεύουμε λιγότερο τελικά ο κόσμος δεν θα αρρωσταίνει με χρόνιες ασθένειες. Ε, χρόνιες ασθένειες είναι πάντα πολύ πιο ακριβές και θα αποφεύγουμε αυτήν την κατάσταση συνήθως. Ελπίζω να απάντησα στα περισσότερα σχόλια που ακούστηκαν. Μέσα στο χρόνο που μου δώσατε, που είχα στη διάθεσή μου. Και μπορώ να το να συζητήσουμε, μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα μετά την... Εντάξει, αυτά για την παρουσίαση και για τη συζήτηση. Προχωρούμε τώρα στην ψηφοφορία. Έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία δύο γνωμοδοτήσεων για δύο διαφορετικά θέματα τα οποία είναι στη μέση διαταξή μα. Ευχαριστούμε την κυρία Λουδοβίκα Μπανφή για την παρουσίασή της και για τα σχόλιά της. Και πάμε στο επόμενο σημείο που είναι η ψηφοφορία. Αν δεν έχετε την ηλεκτρονική σας κάρτα, θα πρέπει να στείλετε κάποιον να την φέρει.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 Χρειαζόμαστε λίγα λεπτά γιατί από εσά δεν έχουν τι κάρτε ξεκινήσουμε. Θα μετρήσουμε και τις ψήφους αυτών που δεν έχουν ηλεκτρονική κάρτα. Λοιπόν, πρώτο σημείο. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και μεταφορά δεδομένων PNR από τις αεροπορικές εταιρείες προς την Αυστραλιανή Υπηρεσία Προστασίας των Συνόρων η κυρία Σόφια Ιντβέλτ Θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια ή ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Μπορώ να είμαι συντομοτάτη, ότι θεωρώ ότι ως εισηγήτρια μπορώ να συνιστήσω την υποστήριξη αυτής της συμφωνίας. Υπάρχουν πολλά ακόμα σημεία τα οποία είναι σημαντικά και πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Αν δούμε όμως τι πετύχαμε, αν λάβουμε υπόψη ότι αυτό αφορά την Αυστραλία ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα να ξέρουν σαν κυρίαρχη χώρα τι θέλουν να ξέρουν από τα άτομα που ταξιδεύουν εκεί πέρα, νομίζω ότι έχουμε επιτύχει ένα αποδεκτό αποτέλεσμα επί τη βάση των κριτηρίων που είχαμε θεσπίσει πέρσι και ως εκ τούτου η σύστασή ω εισηγήτριας είναι να ψηφίσουμε υπέρ με τις κριτικές σκέψεις που υπάρχουν στην αιτιολογική σκέψη. Ευχαριστώ κυρία Ιντεβέλτ. Ο κύριος Άλμπρεχτ είναι έτοιμος να παρουσιάσει την άποψη της μειοψηφίας. Είναι έτσι. Εμείς ως ε, μέλη της Επιτροπής έχουμε πάντα τη δυνατότητα να καταθέσουμε μια έκθεση μειοψηφίας και υπάρχουν ορισμένοι βουλευτές από την ομάδα των Πρασίνων και από την ΚΟΕ οι οποίοι θέλουν να καταθέσουν μια έκθεση μειοψηφίας για να εξηγήσουμε τη στάση που παίρνουμε στην ψηφοφορία κατά τη εκθέση αυτή. Εγώ δεν είμαι πεπισμένο ότι υπάρχουν αποχρόντες λόγοι να υποστηρίξουμε αυτή τη συμφωνία για τα PNR με την Αυστραλία, λαμβάνοντα υπόψη το μεγάλο χρόνο φύλαξη και τα προφίλ τα οποία χρησιμοποιούνται για περαιτέρω έρευνε. Όλα αυτά θα τα εξηγήσουμε στην ε, δήλωσή μα. Επομένω δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Ωραία. Η ψηφοφορία είναι πολύ απλή ψηφίζουμε το σχέδιο σύστασης ως σύνολο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 7 κατά, μία αποχή. Η έκθεση έχει εγκριθεί. Ευχαριστούμε κυρία Ίντφελτ και τώρα πηγαίνουμε στο επόμενο σημείο. Η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Η κυρία Ελέν Φλότρο. Θέλετε να παρουσιάσετε το θέμα αυτό. Όχι. Ωραία. Ψηφίσουμε. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Δεκτή. Τροπολογία 10. Ψήφι υπέρ. Στην επόμενη σελίδα. Κατά. Αποχέ δεκτή. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Για τροπολογία 10. την ψηφοφορία. Πέρασε. Ισοψηφία σημαίνει απόρριψη. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Γιατί νομίζω ότι θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Ελέγχουμε. Άρχεται την ψηφοφορία. Πέρασε. 18-17. Αυτή τη φορά είναι νεκρή. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Αλλά θα ελέγξουμε γιατί δεν σηκώσανε αρκετά χέρια. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα απολύτω, 15-20. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε έλεγχο για 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 29. Όχι. Δεκαεννέα. Όχι. Όχι. Εκπίπτουνε όλες. Πάμε στην 21 κατευθείαν λοιπόν. λέει ο δικός μου κατάλογος, ότι αν εγκριθεί η 3, οι ακόλουθες εκπίπτουν. Πάμε στη 19. 29 δηλαδή λέει ο πρόεδρος. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκριτ. Δεύτερο τμήμα, υπέρ Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 4. Άρχεται. Now closed. 16 against 20 rejected. 34 and 35. 34 και 35 ταυτίζονται. Εκπίπτουν όλες αυτές τις τροπολογίες. 39 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος και πάλι. Άρχεται. Πέρας. 20-16 εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όλες οι, τροπολογίες, οι άλλες τροπολογίες εκπίπτουν. Πάμε στην συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτουν οι υπόλοιπε τροπολογίε αλλά όχι 58. Ψήφι πέτσι 58. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε και πάλι 58. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 58. Πέρασε. Απεριπτέ. Εξήντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος, έλεγχος βεβαίως. Κάνουμε. Άρχεται ο έλεγχος για την εξήντα. περασε 21 21-15. Απορρίπτεται. Σαφώς. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Κάποιες τροπολογίες εκπίπτουν. Πάμε στην 71. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομίζω τουλάχιστον ότι εγκρίνεται έλεγχος ηλεκτρονικός για την 72. Άρχεται. Πέρασε. Για την 72. Χωρίς μικρόφωνο επανάληψης 72 από την αρχή. Άρχεται η ψηφοφορία. Now closed. Πέρας. 24-13 απορρίπτεται και τώρα η τελική ψηφοφορία, το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί, με ηλεκτρονική διαδικασία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας. 35 υπέρ, 2 <clears throat> κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Φλότρο. Προχωρούμε. Στο επόμενο σημείο. Σημείο υπαριθμών 6. I don't see him in the room yet. Όσοι είχατε έρθει για την ψηφοφορία, σας ευχαριστούμε. Καλά ήρθατε στην ψηφοφορία. Θα θέλαμε τώρα όμως ε, όσοι είναι εδώ να σοπάσουν για να περάσουμε στο επόμενο σημείο που αφορά την κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση στην περιοχή της Μεσογείου επαναπροώθηση, επαναγκατάσταση και παρεχόμενη βοήθεια από την Επιτροπή. Θα ακούσουμε μια παρουσίαση του κυρίου Μανσερβίζη, ο οποίος δεν έχει φτάσει ακόμα. Θα κάνουμε λίγα λεπτά διάλειμμα. Μέχρι να έρθει εδώ ο εκπρόσωπος της Επιτροπής 5 λεφτά, 10 λεφτά. 15 λεπτά διάλειμμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι 4 και 4 ακριβώ και είμαστε όλοι εδώ και έτοιμοι. Συνεχίζουμε με τη μέση διάταξη στο σημείο 6, η κατάσταση για τη μετανάστευση στην Μεσόγειο. Επαναπρόθεση, επανεγκατάσταση και βοήθεια που παρέχει η Επιτροπή. Θα ακούσουμε την παρουσίαση του κ. Στέφαν Ματσερβίζη, Γενικός Διευθυντής Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επίτροπος Μάλστρομ, που την είχαμε προσκαλέσει, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα και στέλνει στο πόδι της το Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Στέφανο Μασερβίζη, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Και θα ακούσουμε τον κύριο Μασερβίζη και επειδή θα έχουμε 45 λεφτά στη διάθεσή μας, θα υπάρχει και χρόνος για να γίνει μια κάποια συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θέλω να δώσω κάποιες βασικές πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι απόλυτα καινούριε για σας. Πέραν του θέματος της εκκίνησης του διαλόγου για την κινητικότητα και την ασφάλεια, αλλά μερικά βασικά γεγονότα πρώτα απ' όλα. Η Κομισιόν, όπως ξέρετε, επενδύει σημαντικούς δημοσιονομικούς πόρους για να βοηθήσει αυτή τη διαδικασία μεταρρύθμισης της διαχείρισης των μεταναστών και προσφύγων, να σας δώσω ορισμένα στοιχεία. 75 εκατομμύρια για να βοηθήσουμε τους μετανάστες που αποχωρούν από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3,6 εκατομμύρια για να δημιουργηθεί ένα περιφερειακό πρόγραμμα προστασίας για τα άτομα τα οποία έχουν βρεθεί μετέωρα σε μια περιοχή και θα τα εφαρμόσει αυτά η Πάτη Αρμοστία για τους πρόσφυγες, 7, 10 εκατομμύρια επιπλέον για την Αίγυπτο, Λιβύη και την Ισία για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση μετά από την κρίση και την ε, επαναενσωμάτωση αυτών οι οποίοι δεν μπορούν να γυρίσουν στις χώρες τους και τέλος το λεγόμενο εαρινό πρόγραμμα το οποίο έχει μόλις εγκριθεί 350 εκατομμύρια για τις χώρες της Βόρειας Αφρικής ως πρόσθετα κονδύλια πέραν των κονδυλίων που υπάρχουν ήδη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και για μια πλειάδα στόχων μεταξύ των οποίων και η αντιμετώπιση των προβλημάτων κινητικότητα και μετανάστευσης. Αυτή είναι η πόλη που έχει κινητοποιήσει η Κομισιόν. Δεύτερον, για τους ανθρώπους, για τα θέματα της επανεγκατάστασης. Η υπάτια αποστία έχει ήδη 3.500 ε, άτομα τα οποία είναι ε, ουσιαστικά χαμένα στο χώρο σε διάφορα στρατόπεδα. Η κυρία Μάλστρομ έχει πιέσει να υπάρξουν ενέργειες επανεγκατάστασης. Υπάρχουν 7 κράτη-μέλη που έχουν Ναι, θα λάβει το λόγο στη συνέχεια, κυρία Ναι. Δεν ήξερα αν είπα κάτι λάθος ήδη, λέει ο κύριος Μανσερβίζη. ...408 τόποι επανεγκατάσταση για πρόσφυγες από τη Βόρεια Αφρική. Προφανώς αυτό είναι μια θετική ενέργεια, αλλά δεν επαρκεί. Το είπε και πολλές φορές και η ίδια η Επίτροπος Μάστρομ. Ελπίζω ότι κάποιες από τις 3.083 ε, τοποθεσίες που έχουν προταθεί για συγχρηματοδότηση θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή και πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα θέματα αυτά. Για το κοινό τώρα πρόγραμμα επανεγκατάστασης προς το παρόν είναι μπλοκαρισμένο λόγω μιας διαφωνίας επί της διαδικασίας. Θα ήθελα και εγώ να βοηθήσω να ξεπεραστεί αυτό το, αυτή η εμπλοκή που είναι ακόμα σε πολιτικό επίπεδο είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να βασιστούμε σε αυτό το πρόγραμμα για να οικοδομήσουμε και το μέλλον. Και φυσικά οι προοπτικές για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο βασίζονται σε σημαντικό βαθμό σε αυτά τα οποία προτείνει το Κοινοβούλιο για την τρέχουσα περίοδο. Τώρα, ο αριθμός των ατόμων που έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως μέσω Ισίας και Λιβύης, ξεπέρασαν τις 60.000. Ο αριθμός αυτός η μεγάλη πλειοψηφία τους έφτασε στην Ιταλία και περίπου 3-4.000 στη Μάλτα. Είναι σημαντική αριθμή λοιπόν των ε, προσφύγων αυτών. Η Κομισιόν έχει κινητοποιήσει τις προσπάθειες υποστήριξης από τα κράτη-μέλη, ιδίως με την επιχείρηση Ερμής, Ήταλο και Μινέρβα εξακολουθούν να είναι ε, ενεργές αυτές οι επιχειρήσεις για την περιπολία των υδάτων του Μαρόκου. Η Europol έχει ξεκινήσει τον εντοπισμό πιθανών εγκληματιών. Υπήρξε πρόσθετη χρηματοδοτική υποστήριξη, επίσης και επαφή με τις τυνησιακές αρχές για να εξασφαλίσουμε ότι θα ενταθεί η συνεργασία στη διαχείριση των συνόρων. Για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε περαιτέρω δραστηριότητε και την Frontex τη προσπάθεια του, η Κομισιόν έχει προτείνει, το ξέρετε πολύ καλά, γιατί και εσεί παίξατε ένα κομβικό ρόλο στο εγχείρημα αυτό, πρόσθετα 52 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν εν μέρη εκταμιευθεί και έχουν δοθεί στη Frontex για αυτήν την ε, επιχείρηση. Ο άλλο φορέα, ο ΕΑΣΟ, ο οποίο εργάζεται για τα θέματα παροχή ασύλου, προετοιμάζεται να παίξει ένα ρόλο από τη στιγμή που θα έχουμε φτάσει μια κρίσιμη μάζα, ξέρετε ότι αυτός ο φορέας έχει μόλις δημιουργηθεί, αλλά έχει πολύ καλή θέληση, έχει καλή υποστήριξη από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη και μέχρι το τέλος του έτους η Κομισιόν θα κάνει μια πρόταση για τη δημιουργία του συστήματος Eurosul που θα σημαίνει καλύτερη διαχείριση των συνόρων στο νότιο τμήμα της Μεσογείου. Τελευταίο ε, σημείο, το πιο καινούριο, είναι η κίνηση διαλόγου για την ε, εταιρική σχέση για την κινητικότητα και την ασφάλεια, ε, όπως είχε προναγγελθεί από την Κομισιόν το Μάιο, το είχε ζητήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο. Και εγώ προσωπικά είχα πάει στην Τινησία πριν από δύο εβδομάδες και την περασμένη εβδομάδα στο Μαρόκο και είχα συνομιλίες με τις αρχές και της Τινησίας και του Μαρόκου για να ξεκινήσουμε επίσημα αυτό το διάλογο ο οποίος ε, υποτίθεται ότι θα μας ε, οδηγήσει στη δημιουργία εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια. Ε, στην Τινησία, παρά το γεγονός ότι έχουν εκλογές, ε, ήταν πολύ θερμή απέναντι στην ιδέα. Το ίδιο και στο Μαρόκο, παρότι ε, δεν έχουμε μεγάλη πίεση από το Μαρόκο. Από τις επαγές που είχαμε, τον Υπουργό, που είχαμε τον Υπουργό Εσωτερικών και Εξωτερικών Υποθέσεων και με διάφορους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των συνόρων και την εφαρμογή του νόμου, με το Υπουργείο Εργασίας ε, και με το Υπουργείο που ασχολείται με τις κοινότητες στο εξωτερικό όλοι ε, συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εταιρική σχέση για αυτά τα τρία θέματα ε, μετανάστευση, κινητικότητα και ασφάλεια, δηλαδή ισοτιμία, εφαρμογή του νόμου στη διαχείριση των συνόρων, δημιουργία καλύτερων, ε, καλύτερων συνθηκών για την κινητικότητα των ατόμων, δηλαδή να μπει επιτάπητο η προοπτική μια συμφωνία διευκόλυνση των θεωρήσεων με την Τινησία και το Μαρόκο, με τι δύο αυτέ χώρε, ε, με συμφωνία επανεισδοχή. Πάντα υπάρχει αυτή η συνοδεία τη συμφωνία επανεισδοχή. Είναι κλασική προσέγγιση με πλήρη εκμετάλλευση τη δυνατότητα που μα δίνει η τοπική συνεργασία Σέγγεν και η προώθηση τη νόμιμη μετανάστευση, δηλαδή δημιουργία ενό περιβάλλοντο όπου τα κράτη-μέλη, τα οποία προφανώ είναι οι κύριοι των αριθμών, μπορούν να αποφασίζουν με πιο άτυπο τρόπο για το πώ θα παντρέψουν την προσφορά και τη ζήτηση που συχνά δημιουργεί προβλήματα και απογοητεύσει και στι δύο πλευρέ. Όταν δεν, φτάνουν τα, φτάνουμε τα νούμερα ή όταν ας πούμε, υπάρχει μια προσφορά η οποία δεν γίνεται δεκτή. Αυτοί οι τρει πυλώντε ε, συζητήθηκαν διαμακρών, ο διάλογο έχει ξεκινήσει. Θα κάνουμε μια άλλη συνάντηση και στην Τινησία και στο Μαρόκο πριν το τέλο του 2011 και το μοντέλο μα είναι η εταιρική αυτή σχέση η οποία ε, όπως δημιουργήθηκε και με την Μολδαβία και με την Γεωργία που έχει προχωρήσει αρκετά ε, και δεν θέλουμε αυτή η ασυμμετρία μεταξύ της Ανατολής και του Νότου να συνεχιστεί, να σταματήσει κάποια στιγμή θέλουμε. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις, οι πολύ πρόσφατες. Στο Μαρόκο ήμουνα την Πέμπτη, ε, στην Τινησία την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, όπως σας είπα, η διαδικασία. Θα βοηθήσει, ελπίζω, τις τα κράτη-μέλη που είναι πολύ δραστήρια και ενδιαφέρονται άμεσα, αλλά όλους μας γενικότερα. Ε, γιατί το θέμα του ασύλου, της μετανάστευσης και της ασφάλειας ε, πρέπει να τύχει καλύτερη διαχείριση Αυτά. For your presentation. You made it speedy. Ευχαριστώ, ήσασταν τάχιστος, θα μας βοηθήσει στη μετέπειτα συζήτηση. Γιατί έχουμε μέχρι τις παρατέταρτο προβλέψει αυτό το σημείο και υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να πάρουν το λόγο. Δύο λεφτά έχει ο καθένα to... Δύο λεφτά το πολύ, ούτως ώστε να μιλήσουν όλοι. Γιατί υπάρχουν πολλοί που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κ. Μπουσουτήλ είναι ο πρώτο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον Γενικό Διευθυντή για την εισαγωγή του. Έχω τρει σύντομε ερωτήσει. Καταρχά είπατε ότι 408 άτομα έχουν προσφέρει οι ευρωπαϊκές χώρες για την επανεκατάσταση ατόμων οι οποίοι έχουν κολλήσει στα σύνορα της Τινησίας με τη Λιβύη. Μία αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πήγε σε αυτή την περιοχή στη Σούσα τον Ιούλιο και περίπου 5.000 άτομα είχαν μπλοκαριστεί εκεί εκείνη την εποχή αλλά εξακολουθούν να είναι μπλοκαρισμένοι, κολλημένοι εκεί. Ε, πώς από αυτά τα 400 μέρη που έχουν προταθεί κάνουν κάτι, για αυτά κάνουμε κάτι. Για τις ε, αρχές της Τινησίας μας είπατε ότι προτίθεστε να δημιουργήσετε μια ε, εταιρική σχέση για τη Συμφωνία Κινητικότητας. Υπάρχει όμως πρόοδος με τις αρχές της Τινησίας. Ξεκινήσατε τις συζητήσεις με τις αρχές αυτές. Ξέρω ότι βρίσκονται σε μια δύσκολη προεκλογική περίοδο και αυτό τους απασχολεί κυρίως. Αλλά πέστε μου, υπάρχει μια κάποια πρόοδος στις συνομιλίες. Και για την ΕΑΣΟ, μας είπατε ότι δεν είναι πλήρως λειτουργικός αυτός ο φορέας, αυτή η υπηρεσία. Πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά. Ο κ. Μωράης. Και εγώ θα είμαι πολύ λακωνικός. Καταρχάς, και εγώ ήμουν στην αντιπροσωπεία που πήγε στην Τινησία. Ε, και πέφτει σε αυτούς ένα μεγάλο φορτίο, δυσανάλογο. Τι δεσμεύσει υπάρχουν, τι έχει γίνει. Αυτό ο διάλογο για την εταιρική σχέση βοηθάει τη διαδικασία, έχει προσθέμενη αξία. Περιγράψατε τη διαδικασία, αλλά πώ θα απελευθούν περισσότερα κονδύλια από τα κράτη-μέλη, από αυτά που έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα, για τη Frontex. Μιλήσατε για την επιχείρηση Ερμές πολύ σύντομα. Η ομάδα μου ρωτάει να μάθει ποια είναι η κατάσταση. Γιατί είναι μια κρίσιμη επιχείρηση για να αναλύσουμε ποιος γίνεται δεκτός, ποιος όχι, ειδικά από τη Λαμπεντούζα. Τι ενημέρωση έχετε. Τρίτη ερώτηση, που είναι πολύ μεγάλη σημασία για όλες τις ομάδες. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για την απελευθέρωση του προγράμματος επανεκατάστασης, γιατί από τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο είναι σαφές ότι όλες οι πολιτικές ομάδες ε, το ζητάνε, οι βασικές πολιτικές ομάδες, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, ποιες είναι οι συνθήκες οι ακριβείς όπου τα κράτη-μέλη ε, δέχονται που δέχονται ε, με τα τοπισμένα άτομα ε, με δυσανάλογο όμως τρόπο μπορούν να επωφεληθούν από την οδηγία για την ε, προστασία αυτών των ατόμων. Ε, κυρία Λάτφορντ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ένα σύντομο ερώτημα μονάχα. Ο κύριος Μασερβίζη αναφέρθηκε στο ότι ο του πυλώνας έχει να κάνει με την νόμιμη μετανάστευση. Όπως γνωρίζει, να στα κράτη-μέλη να κάνουν συγκεκριμένε αριθμητικέ προσφορές για νόμιμη μετανάστευση, αλλά υπάρχουν προοπτικές για οποιασδήποτε τέτοιου είδου προσφορές από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει διάλογο σε σχέση με την νόμιμη μετανάστευση στα πλαίσια κάποιων απτών προοπτικών να υπάρξει νομιμοποιημένη μετανάστευση ή όχι. Ή γίνονται όλα αυτά σε ένα κόσμο φαντασιακό. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. για τους 408 οι οποίοι θα μπορούσαν να επανεγκατασταθούν. Είναι μέσα στην ποσόστοση ή έξω από την ποσόστοση. ποσόστοση της δικής μου χώρας ήταν 55 σε, στην ποσόστοση Θα ήταν καλό να ξέρουμε αν οι ευρωπαϊκές χώρες θα αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους ή όχι. Για τη Λιβύη. Το καλοκαίρι του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε μια συμφωνία με τη Λιβύη για την προστασία των συνόρων και υπήρξαν κάποια ποσά τα οποία μεταβιβάστηκαν από την Κομισιόν στη Λιβιακή κυβέρνηση, στη Λιβική κυβέρνηση που ήταν ακόμα ο συνταγματάς Καντάφη. Δεν μας είπατε τίποτα για αυτή τη συμφωνία και τι, αν εφαρμόζεται Μπορείτε να μας πείτε και για την αναθεωρημένη, ανανεωμένη συμφωνία Λιβύης με Ιταλία. Και αν κατάλαβα καλά, το προσωρινό συμβούλιο που έχει την εξουσία στην ε, Λιβύη κατά πόσο εκτελεί περιπολίες στις θάλασσες. Και τέλος για την νόμιμη μετανάστευση. Έχουμε μια, μετανάστε... Έχουμε μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο για τους ε, εποχιακά εργαζόμενους κτλ. Πιστεύω ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες της Βόρειας Αφρικής να ευημερίσουν περισσότερο, θα πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να δείξουν μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με την εποχιακή μετανάστευση. Είναι αυτό το τμήμα της συζήτησης ή όχι. Ο κύριος Ιακολίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μανσερβίζη. Το είπε και ο Διευθυντής. 60.000 άτομα τους εννέα πρώτους μήνες του 2011. Πολύ πολύ στη Σικελία. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στείλει μια αντιπροσωπεία τέλος Νοεμβρίου και θα κάνει και μια, ένα ταξίδι στη Λαμπεντούζα. Ε, μας μίλησατε για τη Λιβύη, ε, είναι πολύ χρήσιμο για την Ιταλία και για το Μαρόκο και για την Τινησία, ούτω ώστε να έχουμε όσο μπορούμε πιο ομαλά νούμερα. Πέρα από το θέμα των προθεσμιών, δηλαδή πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για την ε, συμφωνία, αυτά τα αντισταθμιστικά μέτρα που ανέφερε πολλές φορές ο Μπαρόζο, εκεί ειδικά όπου δέχονται πολλά, πολλούς μετανάστες, Λαμπεντούζα, Σικελία, Λαμπαντερία. Ε? Παντελερία, συγγνώμη. Ε, χρειαζόμαστε απαντήσεις γιατί ε, αυτές οι περιοχές πραγματικά, ε, οι περιοχές έχουν ανάγκη από μια απάντηση. Η κυρία Γκόνς. Δεν ζήτησατε το λόγο. Η κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο διάλογος για την εταιρική σχέση για την κινητικότητα με τις χώρες της, νότης, της Νότιας Μεσογείου είναι πολύ σημαντικός και τον Ιούνιο παρουσιάστηκε μια πρωτοβουλία που μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα. Το πρόβλημα είναι ότι η κατάσταση υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Η... Το γραφείο αυτό για το άσυλο στη Μάλτα δεν λειτουργεί. Στη Μάλτα, στην Ελλάδα, στη Λαμπεδούζα έχουμε τέτοια στρατόπεδα κρατήσεων. και που δεν έχουν καμία σχέση με τις ανθρώπινες αξίες που υπερασπιζόμαστε. και μας μιλάτε για 500 εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα μοιραστούν αυτά τα λεφτά, πώς θα χρησιμοποιηθούν. Έχει γίνει καμία αξιολόγηση, τουλάχιστον εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Ελπίζω να έρθει η Επίτροπος ή τουλάχιστον κάποιος να μας δώσει περισσότερες εξηγήσεις, ούτως ώστε να ξέρουμε λίγο καλύτερα ε, ότι καταρχάς υπάρχουν αυτά τα κονδύλια και τι χρήση θα τους τους επιφυλάσσουμε. Επίσης, ε, ανησυχούμε για αυτά που σημαίνουν στα σύνορα ε, την Ισίας και Λιβύης. Λέτε ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Επανεκατάσταση. Υπάρχουν ε, κονδύλια, υπάρχει ένα ταμείο το οποίο δεν χρησιμοποιείται πρέπει να αποδεσμευτούν αυτά τα κονδύλια. Θα, μπορείτε να, θα μπορούσατε να μου πείτε επίση τι είναι αυτό το Ευρωσούρ. Ευχαριστώ. ο Μούλτερ, λέει Thank you. I can imagine that from Libya we have a lot of refugees. Έχουμε πολλού μετανάστε, αλλά ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που έγιναν μετά την Επανάσταση στην ε, Ισία είναι ότι από την Τινησία είχαμε επίση και ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ήρθαν. Πώς λοιπόν βλέπετε τα πράγματα αυτή τη στιγμή με τους ε, πρόσφυγες από την Τινησία. Ποια είναι τα αποτελέσματα των γεγονότων στην Τινησία, στην Αίγυπτο, στη Συρία. Τι περιμένει η Κομισιόν. Είναι έτοιμη η Κομισιόν, προετοιμάζεται για μια νέα εισρωή προσφύγων. Ευχαριστώ. Αναφέρατε τα νούμερα της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τα, τις χιλιάδες προσφύγων που περιμένουν επανεκατάσταση. Η ΥΠΑ της Αρμοστία επίσης λέει ότι τουλάχιστον 2.000 ε, άτομα από τα μέσα Φεβρουαρίου πνίγηκαν ή πέθαναν στη Μεσόγειο. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά νομίζω ότι η απάντηση που μας έδωσε μέχρι στιγμής δεν είναι ικανοποιητική γιατί μας λέει Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω περισσότερα από αυτά που σας είπα. Δεν συνέβησαν στα ευρωπαϊκά ύδατα. Και από πλευράς Frontex ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Υπενθυμίσατε ότι δίνονται αρκετά κονδύλια για να διαχειριστούμε τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στη Μεσόγειο που υπάρχουν 2.000 νεκροί. Δεδομένου των πολλών πλοίων που κυκλοφορούν στη Μεσόγειο είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε πιο απαιτητικοί. Γιατί η κατάσταση είναι δραματική. Παρότι από τη στιγμή που κατέλαβαν την ε, Τρίπολη βλέπουμε ότι δια της βίας μεταφέρονται άτομα. Εμείς ε, θα πρέπει να απαιτήσουμε να χυθεί απλωτοφώς σε αυτήν την ε, απαράδεκτη κατάσταση. Ε, προβλέπεται η συμφωνία σε εταιρική σχέση για τη Μεσόγειο. Τελειώνω, τελειώνω. Μιλάτε για ένα μικρό πακέτο με ρήτρε για την νόμιμη μετανάσταση, διαχείριση των συνόρων, κατά αποτλέμιση συμφωνίες συμφωνίε επανεισδοχή, μπλα μπλα μπλα. Ε, τέτοια πράγματα έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν στα ανατολικά της Ευρώπης. Ε, έχετε διδαχθεί τίποτα, πώς λειτουργεί, πώς δουλεύει, ειδικά όταν υπάρχουν ισορροπίες, γιατί η Συμφωνία επανεισδεχής είναι το δικαίωμα ε, απέλασης από όλα τα κράτη-μέλη προς τις ενδιαφερόμενες χώρες. Όμως η κινητικότητα και η διευκόλυνση των θεωρήσεων ε, αυτό εξαρτάται από την καλή θέληση των κρατών μελών. Αυτή η έλλειψη ισορροπίας πώς λειτουργεί εκεί που το έχουμε εφαρμόσει. Ε, μια και θέλουμε να πειραματιστούμε με το ίδιο πράγμα στο νότο της Μεσογείου. Της Μεσογείου. Και μια τελευταία παρατήρηση. Οποιοδήποτε παρακολουθεί την ε, προεκλογική εξατία στην Τινησία βλέπει ότι πέρα από τις τεράστιες διαφορές ε, των διαφόρων εκλογικών καταλόγων, του πλουραλισμού κτλ, όλοι, σχεδόν όλοι οι λένε ότι η μεταβατική κυβέρνηση είναι μεταβατική, όλες οι αποφάσεις ε, που θα πάρει θα τις αναθεωρήσουμε όταν δημιουργηθεί νέα συντακτική συνέλευση κτλ. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί απέναντι σε αυτούς τους συνομιλητές μας. Γιατί τώρα οι τινήσοι αρχίζουν, ψάχνονται ακόμα και αρχίζουν να επιλέγουν. Εξάλλου το σχέδιο ε, Jasmine ε, το στυλιτεύουν όλοι οι εκλογικοί κατάλογοι. Για τις συμφωνίες αυτές κινητικότητας λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Η κυρία Άννα Γκόμες. Ευχαριστώ. Ούτω ή άλλω δεν βγαίνουν πολλοί από τη Λιβύη. Οι περισσότεροι Λίβοι που φύγαν προ την Τινησία και στι γειτονικέ χώρε λόγω του πολέμου δεν επέστρεψαν στην Λιβύη. Έχουμε το πρόβλημα των 5.300 που ήταν στην Τινησία και του έχει εντοπίσει η Πατιαρμοστία και είχε πει ότι ήταν είτε τούντες άσυλο είτε πρόσφυγες. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα. Κύριε Μανσερβίζη, πέστε μας τι κάνετε εσείς για να πείσετε τα κρατημέλη να κάνουν περισσότερες προσφορές για να εξασφαλίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Στην ε, Λιβύη είχαμε τουλάχιστον 1.500 ανθρώπους σε ένα στρατόπεδο κοντά στην ε, Τρίπολη. Ίσως υπάρχουν και άλλα στρατόπεδα. Το ενδιαφέρον είναι ότι από τη στιγμή που έπεσε η Τρίπολη στους ε, επαναστάτες δεν πηγαίνουν πια πλοία προς τη Μάλτα ή προς αλλού. Αυτό ε, σημαίνει ότι το χρησιμοποιούσε ο Καντάφη για να εκβιάζει τους δικούς μας. Ε, δεν υπάρχουν άλλα πλοία με πρόσφυγες. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι πρόσφυγες μεν, δεν έχουν χαρακτηριστεί έτσι, αλλά μετανάστες που θέλουν να επαναπατριστούν και για τους οποίους πρέπει να κάνουμε κάτι. Κύριε Μασερβίζη, κάνουμε κάτι μέσω του, της είπα της αρμοστίας για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μπλοκαρισμένοι στη Λιβύη και ε, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι για τις χιλιάδες που πρέπει να επαναπατριστούν από την, ε, όταν απελευθερωθούν από τις φυλακές. Ε, μιλάμε για μισθοφόρους που είναι σε φυλακές της Λιβύης ε, που τους κατηγορούν ότι ήταν ε, μισθοφόροι του Καντάφη και πολλοί θέλουν να πάνε στη χώρα τους πίσω και πρέπει να πάνε να πατήσουν να φύγουν από δηλαδή. Τέλος, τι μπορούμε να κάνουμε για να πείσουμε τα κράτη-μέλη για να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα, το κοινό πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Τι επιχειρήματα χρησιμοποιούν για να μπλοκάρουν αυτό το πρόγραμμα, για να μην τεθεί σε ισχύ. Νομίζω ότι είμαστε σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Αν, α πούμε, υπάρξει μια κρίση στην Αλγερία, Ποιο ξέρει, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί τα πράγματα να δυσκολέψουν πάρα πολύ. Κύριε Σταβάρη. Για την ε, επανεγκατάσταση έχουμε καλά νέα ότι η Επιτροπή να ανέκρινε το πιλωτικό πρόγραμμα για την επανεγκατάσταση και φαντάζομαι θα εγκριθεί και στη συνέχεια και από την Ολομέλεια. Για το μπλοκάρισμα τώρα της ε, συναπόφασης για τα θέματα επανεγκατάστασης, όπως ξέρετε, κύριε Μανσερδίζη, υπήρχε μια πρόταση κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας που κι εσείς είχατε συμμετάσχει σε αυτό το εγχείρημα Εγώ συναντήθηκα με τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις άλλες πολιτικές ομάδες και έχουμε κάνει μια αντιπρόταση να προωθήσουμε την κατεξουσιοδότηση πράξη η οποία ήταν το δύσκολο σημείο για την ε, συναπόφαση είναι μια διαφορά που έχει να κάνει μονάχα με την ανάγκη μιας περαιτέρω συνάντησης για να συμφωνήσουμε για τα θέματα αυτά αλλά δεν έχουμε καμία απάντηση από την Κομισιόν ή από το Συμβούλιο στα ερωτήματα που θέσαμε. Εμείς ξεκινάμε τώρα τις συνομιλίες με την Δανική Προεδρία, η οποία εργάζεται μαζί με την Πολωνική Προεδρία για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Αλλά αυτό πρέπει να λυθεί μέσα στην Πολωνική Προεδρία, αλλιώς θα χάσουμε ένα πλήρη χρόνο θα χάσουμε αλλιώς. Ίσως η Κομισιόν λοιπόν μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσει την αντιπρόταση του Κοινοβουλίου καταρχήν και να μας πει τι, τι θεωρεί ότι ποια είναι η απόψη της για αυτή την πρόταση και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε διάλογο το ταχύτερο δυνατό. Αλλά χρειάζεται πραγματιστική και ταχεία δράση. Λοιπόν, είναι θέμα σαφήνειας. Είναι Δεν είναι μια διαφωνία του Συμβουλίου με το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει κάνει δύο φορές τη δουλειά που έπρεπε να κάνει, πρώτα με τη συναπόφαση και μετά με την αντιπρότασή του. Δύο φορές το Συμβούλιο εκόφευσε σε αυτά τα οποία λέμε. Ελπίζω ότι στο υπόλοιπο της πολιτικής Προεδρίας θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό, αλλά θα ήθελα και τη βοήθεια της Κομισιόν για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά. Κάτι ακόμα το οποίο θέλω να αναφέρω για τα προβλήματα της ε, απόθεσης ορισμένων προσφύγων από την, ε, την, Ισία, από την Ιταλία προς την Ισία Οι Ιταλικές αρχές είπαν ότι αυτό εμπίπτει στη διμερή του συμφωνία. Επομένως θα ήθελα να ξέρω αν η Κομισιόν γνωρίζει αυτή τη συμφωνία και αν θεωρεί ότι αυτή η διμερή συμφωνία εμπίπτει, μάλλον ανταποκρίνεται στις ε, ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και εάν ισχύουν αυτά τα πρότυπα, γιατί υπάρχει αυτή η επαναπρόθεση. Και επίσης για τη Λαμπεδούζα, ποιες είναι οι συνέπειες του γεγονότος ότι έχει θεωρηθεί ασφαλής λιμήν και αν αυτό θα επηρεάσει την ασφάλεια άλλων προσφύγων και ετούτων άσυλο στη Μεσόγειο. Κύριε Μπρόνς, θέλετε να λάβετε το λόγο. Βεβαίως. Μα <clears throat> ότι ο κύριος Κάμερον και ο κύριος Σαρκόζη βομβαρδίζαν τη Λιβύη για να γίνει μια αγγελική και αγαθή χώρα που χαίρεται να ζει κανείς εκεί. Αλλά φαίνεται ότι πολλοί Λίβοι και την Ίση θέλουν να φύγουν και να έρθουν στην Ευρώπη όταν είχαν δικτάτορες και εξακολουθούν όταν έχουν φύγει οι δικτάτορές τους και τους έχουν διώξει, εξακολουθούν θέλουν να έρθουν. Ίσως όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τις πολιτικές συνθήκες. Θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και να μείνουν στην Ευρώπη γιατί θα περνάνε καλύτερα εδώ. Η αρχή της μη επαναπροώθησης είναι ότι δεν πρέπει κάποιος να ξανασταλεί σε μια χώρα η οποία είναι επικίνδυνη. Αν ισχύει αυτή η αρχή, πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους σε επικίνδυνες χώρες. Όταν φέρουμε όλο τον πληθυσμό της Ασίας και της Αφρικής, ώστε να είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο, και η Ευρώπη βουλιάξει, τουλάχιστον θα έχουμε σεβαστεί την αρχή της μη επαναπρόθεσης και αυτό θα είναι η μόνη μας παρηγορία. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπορσελίνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να μιλήσω για την Ιταλία, Λαμπεντούζα και όλα όσα συνέβησαν πριν από λίγους μήνες με την ε, επιχείρηση της ε, αναγκαστικής, ε, του, ε, του, αναγκαστικής, του αναγκαστικού επαναπατρισμού, συγγνώμη, με όλες τις συνέπειες που υπήρχαν. Επίσης το χωριό Μινέο, όπου η Ιταλική κυβέρνηση έφερε ετούντες ασύλου από όλη την Ιταλία. Τους έχει βάλει εκεί πέρα, εδώ αρκετό, και αρκετό καιρό και προσπαθεί, περιμένουμε ας πούμε, να τους αναγνωριστεί το καθεστώς του ετούντα άσυλο. Είμαστε πάρα πολύ αργοί. Στο μεταξύ τους βάζουμε εκεί πέρα, τους ε, φορτώνουμε, τους συσσωρεύουμε. Ποιο έχει την ευθύνη για όλη αυτή, για αυτή την κατάσταση, όταν οι κυβερνήσει δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τέτοιε καταστάσει και απλώ ε, συσσωρεύουν ανθρώπου τον να πάνε στον άλλον. Ευχαριστώ. Πριν δώσουμε ξανά το λόγο στον κύριο Μανσερβίση για να αντιδράσει, η Πολωνική Προεδρία, μήπως θέλει να πάρει το λόγο, η Πολωνική Προεδρία από το Συμβούλιο. Θέλει να συμμετάσχει στη συζήτηση. Έχει την ευκαιρία τώρα. Μετά το Γενικό Διευθυντή θέλω να πάρω το λόγο. Θα είναι ευκολότερο για σας, αλλά όχι για το Γενικό Διευθυντή. Η συζήτηση ήταν πολύ έντονη. Συχνά ούτω ή άλλω έχουμε τέτοιε συζητήσει στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Α δώσω ξανά τον λόγο στον ε, κύριο Μανσερβίζη και μετά θα ακούσουμε και το Συμβούλιο, την Πολωνική Προεδρία δηλαδή. Νομίζω ότι θα χρειαστεί μια ώρα ακόμα. Οπότε, ίσως κάποιες ε, συνομιλίες μπορούν να γίνουν σε διμερές επίπεδο ή με οποιαδήποτε ευκαιρία βρείτε. Αλλά Σέβομαι το χρόνο, το χρόνο σας ε, και τις, τα άλλα θέματα που έχετε να κάνετε. Τώρα το θέμα της επανεγκατάστασης. Από τις 400 τόσες θέσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, είναι κάπου 100 υποθέσεις οι οποίες έχουν προωθήθει. Δεν είναι μεγάλος αριθμός. Γι' αυτό δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Το είπε και η κυρία Μάλστρομ. Και στενοχωριόμαστε ακόμα για το γεγονός ότι όλες οι προτάσεις οι οποίες έχουν σε στόχο να ενισχύσουν την συλλογική λήψη απόφασης για να προωθηθεί η επανεγκατάσταση πέραν του πιλωτικού προγράμματος και χαιρόμαστε που θα λυθεί το πιλωτικό πρόγραμμα παρεθετικά. Όλα αυτά χρειάζονται πολύ χρόνο λόγω των διαθεσμικών θεμάτων που αφορούν σε εφαρμοστικές ή κάτι εξουσιοδότηση πράξης. Κάποια στιγμή, και αυτό λέει και η τελευταία πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπαμε ας αφήσουμε κατά μέρο τα θέματα Τη θεσμική μηχανική και α προχωρήσουμε σε μια πολιτική απόφαση που θα οδηγήσει σε πολιτική συμφωνία. Α χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή την τελευταία ευκαιρία για να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε προ τα πού θα μπορούσαν να πάνε τα πράγματα προς το μέλλον. η Πολωνική Προεδρία. Φυσικά θα πρέπει σε θεσμικό επίπεδο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά, αλλά σε επίπεδο ουσία θέλουμε να συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα για την εξέβρεση μια λύση. Δεν είναι λαμπρά λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία για την Ευρώπη στα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά στην επαναγκατάσταση Εμεί συνεργαζόμαστε με την υπάθεια αρμοστία για του πρόσφυγες, τώρα οι πρόσφυγε βρίσκονται σε διαφορετικέ καταστάσει αυτά που είπε ο κύριος Μπουσουτήλ <clears throat> ευσταθούν τα αριθμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία που συνέλεξα από την υπάτη αρμοστία του ΟΗΕ στην, στην είναι έγκυρα και θα αυξηθούν κατά πάσα πιθανότητα και υπάρχει υποστήριξη του Περιφερειακού Προγράμματος Επανεγκατάστασης που εκτελούμε μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχουν κάποια από αυτά τα άτομα τα οποία μπορούν να φτάσουν στους τελικούς προορισμούς τους. Έχουμε και τη βοήθεια του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών για την υποστήριξη της ε, επανεγκατάστασης ατόμων από την Τινησία. Επίσης αντιμετωπίζουμε όλους αυτούς που έχουν μείνει μετέωροι στη Λιβύη. Εδώ δεν είναι πραγματικά γνωστά. Γνωστό πόσο είναι ο αριθμός αυτών των ανθρώπων και δεν είναι και σταθερός ο αριθμός τους. Πάρα πολλοί οι οποίοι είναι από την Ποσαχάρη Αφρική φοβούνται ότι θα τους θεωρήσουν με μισθοφόρους γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλοί μισθοφόροι. Και υπάρχουν δύο πραγματικότητες στην ε, Λιβύη. Μία είναι η πραγματικότητα της Τρίπολης, μία της Βενγκάζης. Στην περίπτωση της Βενγάζης είχαμε προχωρήσει σε κάποιες συζητήσεις για την ε, διαχείριση των συνόρων και είχαμε στείλει και μια αποστολή εκεί για να υποστηρίξει τις συντονισμένες δράσεις των κρατών μελών. Παραγωγή χάρη για την ε, παροχή προξενικών θεωρήσεων, ώστε να μην έχουμε μια χαοτική πολιτική, αλλά να βασιστούμε σε αυτά τα οποία κάνουν ήδη ορισμένα κράτη-μέλη, όπως η Ουγγαρία ή η Μάλτα. Αλλά η κατάσταση τώρα στην υπόλοιπη Λιβύη δεν είναι ίδια. αυτα όσον αφορά την επανεκατάσταση και για πέστε μου, αυτό αυξάνεται 400 και κάτι παραπλέον. Ε, νομίζω ότι μέχρι σήμερα δεν ισχύει αυτό μέχρι σήμερα πρόκειται για κάποια δέσμευση, πρόκειται για κάποια απόκριση που έγινε σε αυτή την έκκληση για μια ειδική επανεγκατάσταση. Τώρα τι θα γίνει αυτό στην πράξη, στον επόμενο κύκλο θα το δούμε στο τέλος, αλλά μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι, έρχεται επιπλέον. Αυτό είναι ένα στόχος. Now, on the, Και... Τώρα, τι μπορεί να κάνει η, Άζο. Όχι, δεν, είναι, εμείς από τον Ιούνιο είμαστε λειτουργικοί και έχουν γίνει προσλήψεις και όλα αυτά έχουν καλύψει την επιχείρηση στην Βόρειο Ελλάδα όπου γνωρίζετε ότι εκεί έχουμε σημαντική δραστηριότητα, εκεί που προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την απορρόφηση από την Ελλάδα των ετούντων άσυλο. Βεβαίω και η Άζο είναι σε κατάσταση τιμότητα για περαιτέρω ομάδων, όμω α είμαι θα ε, γιατί έχουμε νέους, είναι, είναι τίμο πόλεμοι και ταυτοχρόνως προσπαθούμε να δούμε πώς θα απορροφηθούν οι πόροι που προβλέπονται ούτως ώστε να μπορέσουμε να ε, έχουμε επιχειρησιακή δυνατότητα για να αναλύσουμε την προέλευση, αυτό που λέμε ΕΑΚ, το curriculum, για να μπορέσουμε να δούμε, ε, έντος το βιογραφικό του καθενός, τι ομάδες θα φτιάξουμε ένα κράτος μέλος κλπ. Πάνω κάτω αυτά μπορώ να σας πω και εμείς συνεχίζουμε να πιέζουμε τα κρατη να κάνουν περισσότερα, να τα κάνουν καλύτερα και, και οι η Επίτροπος με από αυτό. Ακόμη δεν τα καταφέραμε παρόλα αυτά, όμως το έργο μας συνεχίζεται. Επίσης, δεύτερο βασικό σημείο, τι θα κάνουμε με την, ε, την Ισία. Αποστολή. Επικεφαλής ήμουν εγώ. για να μην έχουμε γραφειοκρατία. Οπότε, πήγε η Επιτροπή, η Πολωνική Προεδρία, η EIS, η Frontex και η Europol. Οπότε είχαμε μαζί όλο τον κόσμο και οπότε και έτσι ξαναρχίσανε οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις ρυθμίσεις για το έργο της Frontex και επομένως έτσι είπαμε πως θα υπάρχει συγκεκριμένη συνεργασία με την Europol για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Όπω και για το Μαρόκο. Πόσο θα κρατήσει. Ε, θα κρατήσει αρκετά, διότι έτσι δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτά τα οποία γίνονται σε διμερές επίπεδο με τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο όμω θέλουμε είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναδεχθούμε ό,τι θετικό γίνει μέχρι σήμερα. Όμω, δεν ξέρουμε ακόμα τι περιεχόμενο θα έχουν ή έχουν οι συμφωνίες, ξέρουμε μόνο τι μας λένε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και οι τινησιακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι θα τα πούν με την Ιταλία όσον αφορά την επικράτειά τους, την υφαλοκρηπίδα τους, την Ιταλική τέλο πάντων υφαλοκρηπίδα, τα όρια για να δούνε τι γίνεται όσον αφορά με τους μετανάστες, την, την, την διαρροή από τη χώρα τέλο πάντων. Και γι' αυτό και είπαμε να μα δοθούν όλα τα στοιχεία για το κατά πόσο πληρούνται όλε οι προποθέσει στήριξη του διεθνού δικαίου. Όμω ακόμα δεν μα κοινοποίησαν τι γίνεται με τη συμφωνία. Πώ λειτουργεί. Ε, και για να διασταυρώσουμε τι είπαν οι Τινήσοι και τι είπαν οι Ιταλοί. Όμω ε, εκεί προσπαθούμε να επιχειρήσουμε στα όρια τη φαλοκρηπία του κάθε κράτο μέλου τη θαλάσσιας επικράτησης για να δούμε τι θα γίνει. δεν μπορεί με τη μια να δώσουμε μια λύση ούτε εμει ούτε η Frontex. Όλε οι πληροφορίε συγκλίνουν προ αυτό τώρα όσον αφορά τη συμφωνία με τη Λιβύη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κλείσει κάποια συμφωνία με τη χώρα. Όμω έχουμε ε, μια κοινή δήλωση, τέλο πάντων μνημόνιο, οτιδήποτε, όπω θέλετε πέστε το, ούτω ώστε να έχουμε τη διαχείριση τη διάβαση των συνόρων στα σύνορα στην Νότια Μεσόγειο και έτσι και εκεί να καταπολεμήσουμε την παρόμοια διακίνηση ανθρώπων. Βέβαια τα πράγματα χειροτέρεψαν από κάποια στιγμή ε, γιατί το καθώς Καντάφη πίεζε τον κόσμο, του εκβίαζε να φύγουν. Και με το που έπεσε ο Καντάφη σταμάτησε αυτό. Οπότε φεύγουν μόνο οι πιστοί του Καντάφη. Και έχουμε αυτή την κοινή δήλωση που υπερήχε και οικονομική ρήτρα, η οποία δεν εφαρμόστηκε γιατί υποτίθεται ότι θα βοηθούσε τη Λιβύη να διαχειριστεί την κατάσταση καλύτερα, να αναμπεί στον Ευρωπαϊκό Παρανομαστή. Οπότε τώρα ξαναγυρίσαμε στο Α, ό,τι προβλεπόταν σε αρχή για την Βόρεια Αφρική και είπαμε ότι στη διάθεση των της λιβικών αρχών θα είμαστε εμείς για να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά το είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ποιο. Τι θα γίνει με τους υποσαχάριους που βρίσκονται εκεί, τι θα γίνει με τους εκεί εργαζόμενους, γιατί η λιβική ε, οικονομία δεν μπορεί να ορθοποδήσει χωρίς τους ξένους. Όλα αυτά επομένω θα πρέπει να τα δούμε στην πράξη όσον αφορά την εταιρική σχέση με τη χώρα. Ναι, αυτό θέλουμε να διχειριστούμε, τη διάβαση των συνόρων, την πτυχή ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης για τα σύνορα, για τις μαφίες, για τη διακίνηση των ανθρώπων, την παράνομη και μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά και στην Τινησία, όπως και στο Μαρόκο, οι αρχές ενδιαφέρονται να αρχίσουν τις συνομιλίες με Europol και Frontex και έτσι να μπορέσουν να συνεργαστούν μαζί μας, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Υπάρχει τώρα έλλειψη ισορροπίας μεταξύ επανεισδοχής, και τις σχετικές διευκολύνσεις. Και προσωπικά, όταν παρουσίασα την έκθεση για την εφαρμογή της επαναπροώθησης και των σχετικών συμφωνιών, είπαμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία και ταυτόχρονα να έχουμε ως μόχλευση διευκολύνσεις ιστορίες διαβατηρίων. Έχουμε με τη μία χώρα, έχουμε την άλλη, οπότε όταν εμπλοκή στις συνομιλίες και προσπαθήσαμε να κάνουμε το παζάρι. Δηλαδή να διευκολύνουμε τις βίζες και ταυτόχρονα κάποια μέτρα που να μην είναι à Γιατί είπαμε την νέα συμφωνία ότι τα ίδια θα ισχύσουν για όλους. Επομένως, η διευκόλυνση εισόδου θα ισχύει για όλους και όχι μόνο για εκείνου. που θέλουν. Και η συμφωνία επανεισδοχής και λοιπά θα ισχύει πάλι για όλους. Επομένως, έχουμε θετική εμπειρία από τη δράση μας εις Ανατολάς και το κάνουμε το ίδιο και εδώ και τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε για την νόμιμη μετανάστευση, την μπλε κάρτα, την οδηγία για του ε, εργοδότε, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα γίνεται η εκμετάλλευση των λαθρομεταναστών εργασιακά, κάτι το οποίο συνδέεται και με την παραμοδιακίνηση ανθρώπων. Και αυτό συνδέεται και με την γεννητικότητα των σπουδαστών, των φοιτητών, των ερευνητών. Έχουμε, έχουμε πολλά να κάνουμε. Οπότε όσον αφορά τις άδειε εργασία αυτό παραμένει εθνική αρμοδιότητα, κρατική αρμοδιότητα. Αλλά στην εταιρική συμφωνία με τη Μολδαβία τι κάναμε. Και έτσι προσπάθησαμε να δούμε τι, τι αποφάσεις ελήφθησαν και τι κοινωτικές αποφάσεις ελήφθησαν ούτως ώστε να ζυγιστεί η προσφορά με τη ζήτηση. Και είχαμε 15 χώρες μέλη που μπήκαν σε αυτό το παιχνίδι. Όμως άλλαξαν πολλά επί τη βάση αυτού και άρα αυτό θα πρέπει να μπει στο τραπέζι καθαρά να συζητηθεί από του υπουργούς απασχόληση των ΜΕΝ και των ΔΕ και αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν, δεν προβλέπεται. Παρακάτω. Για το θέμα της αρρωγής της όλης περιοχής και το γίνεται στη Λαμπεντούζα που βέβαια ξέρουμε τι σημαίνει, τι συμβαίνει. Είπαμε ότι πια δεν είναι ασφαλής λιμένας. Κατεστράφησαν οι υποδομές εκεί, οπότε οι Ιταλικές αρχές τώρα έχουν το λόγο. Γιατί χρησιμοποιούσαμε τη Λαμπεντούσα γιατί ήταν κοντά. Και τώρα μεταξύ νησίας και Σικελίας δεν υπάρχει Λαμπεντούζα, μεγάλη απόσταση. Και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και είπαμε στους Ιταλούς να μας εξηγήσουν τι προτίθενται να κάνουν. Απλά να μας πούνε, γιατί βρίσκονται ακόμη πιο στριμωγμένοι. Μάλλον αυτοί χρειάζονται τώρα βοήθεια. Άρα πρέπει τώρα να μας πούν τι κάνουν, τι προτίθενται να κάνουν. Έχουν διεθνές καθήκον. Είμαι σίγουρος ότι κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά είναι πολύ στριμωγμένοι. Οπότε... Μηνέο. Προχωρούν οι συνομιλίες με την Ιταλία. Για να δούμε και εκεί τι θα κάνουν. Όμως, ακόμα δεν έχω στοιχεία για να σας πω. Κατά πόσο έχουν παραβιάσει των δικαιωμάτων. Όχι μέχρι σήμερα. Οπότε, θα γίνει και κάποια αποστολή. Οπότε και θα εξετάσουμε το τι έγινε ή στο μηνέα. Πάντως μέχρι σήμερα τα όσα εκεί γίνονται και στα διεθνή ύδατα και τα όσα μας αναφέρουν δείχνουν ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, αλλά όχι, δεν συνιστά κρίση όπως στην Ελλάδα παρόλα αυτά όμως. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα δούμε. Φυσικά εξαρτώμεθα από αυτά που μας λέει η Ιταλία. για τη χρήση τη οδηγία για την προσωρινή προστασία. Δεν τη χρησιμοποιούμε αυτή την οδηγία. Τελεία. Μπορούμε να συζητήσουμε το γιατί. Αλλά δεν χρησιμοποιείται αυτή η οδηγία γιατί κανένα δεν θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Ίσως πρέπει να το συζητήσουμε για να δούμε είναι χρήσιμη, μήπως πρέπει να τη μεταρρυθμίσουμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και το, 73, το άρθρο 73α, το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε, πρέπει να προβληματιστούμε. Πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε καλύτερα με βάση την εμπειρία που έχουμε. Αλλά αυτό είναι τμήμα μιας ευρύτερης συζήτησης για την αλληλεγγύη. Υπάρχουν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες πρακτικές, καλές πρακτικές, αλλά το να περάσουν αυτά και να γίνουν νομοθεσία, δεν έχουμε φτάσει εκεί. Για τους πνιγμένους. Είναι ένα τρομακτικό δράμα, αλλά δεν έχουμε αποδείξεις που να μας πείθουν ότι πέρα από το πραγματικό δράμα που συνδέεται με τα κακά σκάφη, που τα εκμεταλλεύονται τα εγκληματικά δίκτυα ή κάποιες κυβερνήσεις, πρέπει να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα ε, είναι απόρρια πολέμου, δύσκολων καταστάσεων σε χώρες και ανθρώπων που θέλουν να φύγουν από αυτές τις καταστάσεις. Το θέμα είναι πώς να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά τις προφορίες που συγκεντρώνουμε μέσα από τις κοινέ επιχειρήσεις, joint operations, που είναι συχνά επιχειρήσεις ε, της Frontex, αλλά που κάνει αυτό που ζητάει το κράτος υποδοχής. Οι επιχειρήσεις ε, της Frontex, λοιπόν, κάνει ανάλυση κινδύνου στη Μεσόγειο, ε, κάνει μία, ένα screening, αλλά δεν κινητοποιούνται πολλά κονδύλια. Οι Ιταλικές αρχές όταν υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα από τις Ιταλικές Αρχές πρώτη Frontex, η Frontex κινητοποιείται, αλλά ε, απόκειται στις Ιταλικές Αρχές. Πρέπει να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Να χυθεί το φως. Αυτό κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια στυλιτεύοντας και βάζοντας το σκάνι του κατηγορούμενου τα κρατη Κάνουμε ό,τι μπορούμε στη δύσκολη αυτή κατάσταση. Μερικές φορές, λέει η κυρία Φλότ, υπάρχουν και επιζώντες από αυτά τα σκάφη. Ε, δώσαν συνεντεύξεις για να δούμε τι, ποια είναι η εμπειρία τους. Το ξέρω, το ξέρω. Ούτως ή άλλως ε, το συζητάμε αυτό το θέμα με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη για να καταλάβουμε αν... τι συμβαίνει. Εμείς στη Frontex όμως δεν έχουμε επιχειρησιακό δυναμικό για να κάνουμε έρευνες εμείς οι ίδιοι. Περιμένουμε ε, από, τα κράτη-μέλη να μας δώσουν πληροφορίες, να μας υποβάλουν εκθέσεις. Όσες περισσότερες πληροφορίες, τόσο καλύτερα. Ε, μπορούμε να ζητάμε πληροφορίες από τα κράτη-μέλη και από την ε, ύπατη αρμοστία. Επίσης, μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο που λειτουργεί η Frontex, ούτως ώστε να μην σεβόμαστε απλώς τα ανθρώπινα δικαιώματα με παθητικό τρόπο, αλλά ούτως ώστε να είμαστε εξοπλισμένοι για να λειτουργούμε πιο ενεργητικά πιο δραστήρια. Συλλέγουμε πληροφορίες και μαζεύουμε εμπειρία. Ε, προσπαθούμε να αρχίσουμε το φως, ε, συνεργαζόμενοι με τα κράτη-μέλη, με τις ε, διεθνείς οργανώσεις, με, τους μη κυβερνητικούς, ε, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και με τις τοπικές αρχές, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το πλαίσιο Τη κινητικότητα μετανάστευση και ασφάλεια θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο πιο πλήρε ούτω ώστε να δούμε την κατάσταση και από τη μία και από την άλλη όχθη τη Μεσογείου. Η Eurosur θα κάνουμε μια νομοθετική πρόταση στο τέλο του 2011, το Δεκέμβριο. Ε, είναι ένα σύστημα για να συλλέξουμε όλε τι πληροφορίε από όλε τι διαφορετικέ αρχέ, είτε από την αστυνομία, από τις ε, αρχές εποπτείας της θάλασσας, ε, ε, από τις αρχές δηλαδή που ελέγχουν τις μεταναστευτικές ροές, τις παράνομες μεταναστευτικές ώρες, τα παράνομα εμπορεύματα, το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών και των όπλων. Έχουμε διακίνηση σε πραγματικό χρόνο πληροφοριών. Τι συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες. Ορισμένα κράτη-μέλη είναι πολύ καλά εξοπλισμένα. Πήγα στη Βαλένθια στα γραφεία της Guardia Civil και εκεί είδα ότι πραγματικά έχουν προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το σύστημα συλλογής πληροφοριών. Έκανα σχετικές συζητήσει και με το Μαρόκο και με την Τινησία ούτω ώστε να συμμετάσχουν σε αυτό το σύστημα για να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται για δικά μα και δικά του σύνορα αλλά είναι κοινή πρόκληση ούτω ώστε να σταματήσουμε τους, ε, λαθρέμπορου. Στο μεταξύ, μην ξεχνάμε ότι πνίγηκαν και 2.000 άνθρωποι στη Μεσόγειο. Ε, υπάρχουν πραγματικά εγκληματικά δίκτυα τα οποία δραστηριοποιούνται. Αυτά τα θέματα θα τα αναλάβει η Eurosur, θα δημιουργηθεί τις επόμενες Δεν Έχω πολύ χρόνο για να απαντήσω σε όλα, αλλά είμαι στη διάθεσή σα βεβαίω. Αντίθετα, κύριε Μασεβίζη, σας ευ... εμείς σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειές σας. Μας δώσατε όσο να τον πιο πλήρε ε, απαντήσεις. Πριν... Πριν κλείσουμε όμω τώρα, για να δούμε τώρα, μήπω η Πολωνική Προεδρία θέλει να πάρει τη σκητάλη. Σα παρακαλώ να είστε όσο πιο σύντομο γίνεται, διότι δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε για το τελευταίο πιάτο τη σημερινή συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η εκπρόσωπο Προεδρία. Θα είμαι ναι, όσο γίνεται πιο σύντομη. Διότι όσον αφορά το σύνολο της Μεσογείου, η Προεδρία και το Συμβούλιο γενικότερα είμαστε στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλα αυτά τα διαδήματα, για όλα αυτά τα μέτρα και όλες τις προσπάθειες. Και έχουμε άλλωστε και τη δεδομένες τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Ιουνίου. Έχουμε επίση αυτέ τι πρόσφατε παρεκκλήσει Μαρόκου Τινησία και οι αποστολέ που έγιναν εκεί μα ικανοποίησαν πλήρω. Επίση, θέλουμε να δοθεί συνέχεια ή στι προσπάθειε που ο κ. Μανσεβίτση μα εξήγησε Όντω, ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τι εταιρικέ σχέσεις που έχουμε αναπτύξει, γιατί θίγει για αυτό το θέμα και ξέρετε, ε, συνήθω αυτού του είδου οι συμφωνίε έχουν να κάνουν με θεωρήσεις διαβατηρίων, επανεισδοχή, επαναπροώθηση κλπ. Τέτοιου είδους συμφωνίες, αυτές οι συμφωνίες κινητικότητας όπως ονομάζονται. Και Προσπαθούμε να έχουμε γεωγραφική ισορροπία. Και ελπίζουμε ότι θα το πετύχουμε. Τόσο αφορά τα προγράμματα της επανεγκατάστασης. Ε, συνεχίζουμε το έργο της Ουγγρικής Προεδρίας. Και προσπαθούμε να ξεπεράσουμε κάποια νομικά κολλήματα που υπήρχαν ασχολείται η νομική υπηρεσία. Έδωσε το πράσινο φω για την Ουγγρική πρόταση. Βεβαίω και εμεί θα πάρουμε τη σκητάλη και θα συνεχίσουμε επί τη βάση των όσων προτείνεται και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν. Thank you. Ο πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μανσερβίζη, θέλετε να κάνετε κάποια τελευταία σχόλια. Εάν όχι, σα ευχαριστώ τα μάτια. Κύριε Ταβάρη, παρακαλώ σύντομα προς την Προεδρία, την Πολωνική Προεδρία. Έχετε ήδη αναλύσει την αντιπρόταση του Κοινοβουλίου. Την έχετε ελέγξει μέσω της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου για μια αξιολόγηση. Η πρόταση αυτή είναι υπό εξέταση. Ελπίζω ότι στις 20 του μηνός θα μπορέσω να σας πω όταν θα γίνει η ακρόαση για το άσυλο και την επανεγκατάσταση. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ σύντομα αυτά που είπατε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μανσερβίση. Σας ευχαριστώ που δώσατε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάθεσης. Yes. We shouldn't be... Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε. Σας υπενθυμίζω ότι μετά από το θέμα αυτό έχουμε την συνεδρίαση των συν των ιστών. Το... Την απογευματινή Όχι τώρα. Τώρα έχουμε ένα θέμα στην ημερησία διάταξη. Το 7 συγκεκριμένα. Απλώς σας υπενθυμίζω τη σημασία που έχει ο χρόνος. 7. Ευρωπαϊκό έτος πολιτών. Παρακαλώ. Όσοι μείνουν στην αίθουσα παρακαλώ να μην φωνασκείτε. Όσοι θέλετε να φύγετε να το, να το πράξετε ηρέμος και ησύχως. Ευρωπαϊκό έτος πολιτών 2013. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαν στόχο να θεσπίσει το 2013 ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών <clears throat> για να εστιάσουμε στα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορεί επίσης η άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών να βρίσκεται στο κέντρο της συνέχεια διάταξής μας. Αυτό το ευρωπαϊκό έτος λοιπόν θα αυξήσει την άσκηση των δικαιωμάτων που συνάπτονται με την ευρωπαϊκή υπηκότητα και ιδίως το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Οκτώβριο του 2011 η Επιτρόπη Λίμπα ε, επιφόρησε την κυρία Παπαδοπούλου ως εισηγήτρια για το θέμα αυτό, αλλά προηγουμένως θα ακούσουμε την άποψη από την κυρία Βαντερστίν, η οποία είναι γενική Διευθυντή της Γενική Γενικής Επικοινωνία Επικοινωνίας της Κομισιόν και η οποία θα μας παρουσιάσει το περιεχόμενο της πρόταση της Κομισιόν και μετά ο κύριος Γιαζίνσκι, ο οποίος εκπροσωπεί την Πολωνική Προεδρία, θα λάβει το λόγο και τέλος η εισηγήτριά μας και τα μέλη τα οποία θα θέλουν να λάβουν το λόγο. Καταρχήν ο κύριος Βαταστίν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, στο ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2009, το κοινοβούλιο σας ζήτησε από την Κομισιόν να θεωρήσει το έτος, να κηρύξει το έτος 2013 ως το έτος της Ευρωπαϊκής Υπηκότητος, ώστε να δοθεί απαραίτητη όθηση για τη συζήτηση σε σχέση με τη συζήτηση για τα θέματα υπηκότητας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Έτσι να μπορούν να ενημερωθούν οι πολίτε, ιδίω εν των νέων διατάξεων, αυτέ οι οποίε έχουν ενσωματωθεί στην συνθήκη τη Λισαβόνα. We believe time... Θεωρούμε δε ότι υπό την σημερινή συγκυρία της χρηματοοικονομικής κρίσης το ευρωπαϊκό έτος ε, του Ευρωπαϊκού Πολίτη είναι μια πρωτοβουλία πάρα πολύ σημαντική. Διότι, όπως προαναφέρατε Πρόεδρε, είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι πολίτες Ένωση για τα δικαιώματά τους, αλλά επίσης και για τα προνόμια των οποίων απολάβουν ως πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να τραβήξουμε τους πολίτες για να εμπλεκούν περισσότερο στο πολιτικό γίγνεσθε για το ευρωπαϊκό όραμα. Και οι φετινές ανακοινώσει αλλά και τα όσα θα κάνουμε για κοινωνία το 2013 αποτελούν πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία ούτως ώστε να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε για τις επόμενες εκλογές του 2014. Ο πρόεδρος Μπαρόσο ξεκαθάρισε ότι ο λόγος ύπαρξης της ε, Ευρώπης είναι το να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να γίνουν ισχυρότεροι. Η δε σημερινή χρηματοοικονομική συγκυρία είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία της Ευρώπης. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ότι μαστεί στην Ευρώπη μια κρίση εμπιστοσύνης. Ακριβώ όπω είπε στην ομιλία το Πρόεδρου σε σχέση με την κατάσταση τη Ένωση. Εδώ ενώπιον του Κοινοβουλίου σα στι 28 Σεπτεμβρίου. με το νοσοκομείο για κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρο, εμεί ε, θεσπίσαμε και συμφωνήσαμε πάνω σε έναν χάρτη πορεία, ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το ε, πρόγραμμα των πέντε σημείων και να σπάσει αυτό ο φαύλο κύκλο τη αβεβαιότητα όσον αφορά το κρατικό χρέο και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε αηφορία αλλά και ανάπτυξη. Αυτό το πρόγραμμα το παρουσίασε ο πρόεδρο Μπαρόσο την περασμένη εβδομάδα. η γη στο Κοινοβούλιο και επίσης θα το παρουσιάσει και την επομένη Κυριακή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίσης, είμαι θα ότι ε, τέτοιες ώρες, ώρες κρίσης, το ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν, να γίνουν πιο ισχυροί οι πολίτες, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ζωτική σημασία οι πολίτες της Ένωσης όχι μόνο να στηρίξουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται σε επίπεδο Ένωσης, αλλά επίσης θα πρέπει και αυτοί να εμπλακούν. Εάν δε εξετάσουμε τα αποτελέσματα της στατιστικής του Ευρωβαρομέτρου, εάν εξετάσουμε τι απάντησε ο κόσμος το ερώτημα τι σημαίνει η Ένωση για τους Ευρωπαίους θα επιστώσει το 45% των απαντήσεων ήταν ότι οι Ευρωπαίοι συνεχώς συσχετίζουν με την Ευρώπη την ελευθερία της ε, διακίνησης για να ταξιδέψουν, ε, να δουλέψουν και να σπουδάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτός ο συνειρμός ακολουθείται από το 37% των απαντήσεων που είπαν ότι συσχετίσουν την Ευρώπη με το κοινό νόμισμα, το ευρώ. Επίση, οι πολίτε της Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι η ελευθερία διακίνηση είναι πάρα πολύ βασικό δικαίωμα το οποίο είναι άμεσα συνδεόμενο με την ιδιότητα του πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει αυτή, αυτό το, το, συσχετισμό των ιδιών να τον εκμεταλλευτούμε και έτσι να αναβαθμίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την καθημερινή πρακτική τους εμπειρία να τους δείξουμε τι πάνε να πει, να είναι κανείς πολίτης τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Χρονιά επομένω των Ευρωπαίων πολιτών πρόκειται να μα δώσει μια χρυσή ευκαιρία για να μπορέσουμε να καταδείξουμε ότι είναι ψηλή μας προτεραιότητα, βασική προτεραιότητα ο κόσμος και επίση να τον εξηγήσουμε και να αποδείξουμε πόσο σημαντική είναι όσον αφορά την ιδιότητά του ω ψηφοφόρων για τι ευρωεκλογέ, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η χρονιά, το 2013, επίτηδε εξελέγει και και κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό θα γίνει ακριβώ ένα χρόνο πριν τι εκλογέ του 2014. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία που θα μας δοθεί, ώστε να κινητοποιήσουμε τις εκλογές. Πρόκειται επίσης για την 20η επέτειο της θέσπισης της ιδιότητας του Ευρωπαϊκού Πολίτη, όπως αυτή κατοχυρώθηκε από τη συνέχεια του Μάστερ επίσης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, για να ρίξουμε μια ματιά στο ποιοι θα μπορούσαν οι στόχοι της χρονιάς του Ευρωπαϊκού Πολίτη. Θέλουμε να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματά τους οι Ευρωπαίοι πολίτε, και την ελευθερία διακίνηση βασικά και να τους πληροφορήσουμε. Η πρότασή μας θέλει να υπάρχει περισσότερη συνειδητοποίηση και έτσι να μπορούν εκείνοι να ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διακίνηση, την διαμονή, την ελεύθερη, οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την αίσθηση του ανήκειν. Να αναβαθμιστεί αυτή η αίσθηση. Και το σίγουρο είναι ότι με περισσότερη ελεύθερη διακίνηση των πολιτών πρόκειται να ωφεληθεί άμεσα η ενιαία αγορά που με τη σειρά του αυτό το φαινόμενο θα οδηγήσει σε καταγύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Το 2013 πρόκειται να τονωθεί επίση ο διάλογο, η προβληματική όσον αφορά το πόσο ωφελεί να είναι κανεί πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. The European of Citizens will be... Αυτή η χρονιά το Ευρωπαϊκό πολίτη πρόκειται να τύχει διαχείριση όσον αφορά την επικοινωνία. Και το κατευθυνόμενο όμω επίση θα έχουμε συμμάχου όλους τους εταίρους μας και όλοι θα πρέπει αποτελεσματικά να εμπλακούν. Να εμπλακούν τόσο ώστε να υπάρξει συνεργασία όλων με όλους. Στρατηγική εταίρη μας όσον αφορά αυτή την εκστρατεία πρέπει να είναι σε νοσιακό επίπεδο τα θεσμικά όργανα. Αυτό ήδη έχει τονιστεί στην διοργανική διαθεσμική ομάδα όταν έγινε η ενημέρωση, γιατί εκεί είπαμε ότι Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπούνται. Στην ομάδα εκείνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκάλεσε όλα τα θεσμικά όργανα να κατεβάσουν συγκεκριμένε προτάσει. Και επίση αυτή η πρωτοβουλία να μπορέσει να οδηγήσει σε μια πετυχημένη χρονιά του Ευρωπαίου πολίτη και η βασική εμπλεκόμενη θα είναι στην πράξη τα ενημερωτικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά επίση και οι αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή ή στα κράτη-μέλη. Πρόκειται να καταδραματίσουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και πρόκειται από κοινού να διοργανώσουν ένα σωρό εκδηλώσει. Οι εθνικέ κυβερνήσει αλλά και η κοινωνία των πολιτών και οι φορεί διάφοροι, τα διάφορα δίκτυα θα πρέπει να εμπλακούν οπωσδήποτε. Ο πλευρά τώρα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εμεί θα προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε κάποιο είδου συμπληρωματικέ πρωτοβουλίε με βάση του δικού μα οικονομικού πόρου. Και πρόκειται αυτή μα την εκστρατεία να την απευθύνουμε στον κόσμο γενικά, στο κοινό, αλλά επίση να δούμε και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που χρειάζεται, ώστε το, τα μηνύματα να περάσουν και να διαδοθούν. Εκείνοι οποίοι για πρώτη φορά ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές το 2014, εκείνοι, εκείνοι θα πρέπει να αποτελέσουν στόχο της ενημερωτικής εκστρατείας και θα πρέπει εδώ να τους εστιάσουμε καλύτερα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα κατεβούν να ψηφίσουν. Στατιστικά, οι γυναίκες, οι νέοι και οι λιγότερο μορφωμένοι χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. και έχουμε προτείνει σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ανάληψη δράση. Με ενημερωτικέ εκστρατείε, με την ε, με μέσω τη παιδείας, τη εκπαίδευση, με την ανταλλαγή εμπειριών, ούτως ώστε να αναλυθούν τα, τα, τα υπέρ, τα προνόμια της ελεύθερη διαμονή, τη ελεύθερη διακίνηση. του να είναι κανεί τελικά όλης Ευρωπαϊκή επίση. Θα πρέπει τις υπάρχοντες πλατφόρμες εργασίας να τις ε, χρησιμοποιήσουμε τόσο ώστε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή των πολιτών και έτσι να μπορέσουν αυτοί να, να, να, αξιοποιήσουν ε, και στην πράξη τα δικαιώματά τους και επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και πώς θα χρησιμοποιήσουμε και εκείνη την διαδικτυακή πύλη που αφορά τους πολίτες και την ενημέρωση από την Κομισιόν σαν διάβολος ενημέρωσης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής Λίμπε, Η Κομισιόν με ανυπομονησία θέλει να συζητήσει αυτή την πρόταση μαζί σας. Να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Και μην αμφιβάλλετε ότι θα συνομιλήσουμε μαζί σας, ούτω ώστε να αξιοποιήσουμε αυτή τη χρονιά και το Κοινοβούλιο θα είναι σημαντικός εταίρος, σημαντικός συνομιλητής ε, της Κομισιόν για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Γιαζίνσκι από την Πολωνική Προεδρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ. Ακούστε, έχω ένα σύντομο μήνυμα από την Πολωνική Προεδρία θα είναι πολύ δύσκολο να πούμε όχι σε μια τέτοια υπέροχη πρόταση. Είναι ένα θαυμάσιο κείμενο. Θα υπάρχει καλή διάθεση. Θα το προτείνουμε στι αντιπροσωπείες το συντομότερο δυνατόν. Και για να τα πω και συγκεκριμένα, έχουμε κανονίσει σχεδόν τις ε, ημερομηνίες. Ε, σε τρεις ε, εβδομάδες η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τώρα ασχολούμαστε με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, εν συνεχεία θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ελπίζω σε τρεις εβδομάδε να είμαστε σε θέση να εγκύψουμε σε αυτό το φάκελο. Δεν μπορώ βεβαίως να προδικάσω τη θέση των κρατών μελών, αλλά ελπίζω ότι αυτό το θέμα θα προχωρήσει και το Συμβούλιο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θετικά και το τελευταίο από μένα. Εμείς από, πλευρά, από πλευράς Πολωνικής ε, Προεδρίας πιστεύει, πιστεύουμε ότι η ε, ελευθερία κινήσεων είναι από τις πιο σημαντικές αρχές, δεν πρέπει να την υποτιμούμε και θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε το κείμενο. Ευχαριστώ που ήσασταν σύντομος. Η εισηγήτρια, κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι είναι ενθουσιασμένη και η Πολωνική Προεδρία και ο Γενικός Διευθυντής. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που είμαι εισηγήτρια για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Πιστεύω ότι πολλοί από τους συναδέλφους μου Λένε συχνά ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος πολίτης, σε τι μεταφράζεται αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστούμε, ούτω ώστε να διευκολύνουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, να μετακινηθούν και να εγκατασταθούν ελεύθερα όπου θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνοντάς τους ότι μπορούν ε, να ενημερωθούν εύκολα για τα ε, δικαιώματά τους. Αυτό το προτινόμενο έτος ε, βασίζεται στην έκθεση αυτή του 2010 με τίτλο «Διαλύοντας τα εμπόδια για τα δικαιώματα των πολιτών» και ο σκοπό έχει να φύγουν τα εμπόδια που παραμένουν εδώ και χρόνια και που εμποδίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών. Πριν από δύο χρόνια, 11,9 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών ζούσαν σε άλλο κράτο μέλο. Αυτό το νούμερο θα αυξάνεται και αυξάνεται σε στιγμέ κρίση. Βλέπουμε πολλού νέου απόφοιτου πανεπιστημίων ε, προσπαθούν να βρουν δουλειά σε ένα άλλο κράτο μέλο από τη χώρα του. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι καλό ότι άκουσε το ψήφισμά μας στις 15 ε, Οκτωβρίου το 2010 και τώρα ε, μας έκανε αυτή την ε, ενδιαφέρουσα πρόταση. Στην έκθεσή μου θα μιλήσω για θέματα όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους να εργαστούν και να διαμείνουν ελεύθερα στην επικράτεια ενός άλλου κρατούς μέλος, την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατόμων, ανεξάρτητα από την φυλή ή την εθνική προέλευση σε διάφορες περιοχές της Ένωσης, σε ό,τι αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, την ε, την ε, υγειονομική περίθαλψη, την πρόσβαση σε αγαθά και σε υπηρεσίες. Το δικαίωμα επίσης στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες και στα έγγραφα, την ανάγκη ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και τα δικαιώματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαβίου μάθησης. Θα συζητήσουμε αυτό το φάκελο εν ευθέτω χρόνο έχουμε αυτή την τύχη πριν από τις ε, ευρωπαϊκές εκλογές του 2014. Είναι κατάλληλη στιγμή για να ενθαρρύνουν τους Ευρωπαίους πολίτες να συνεισφέρουν, να συμμετάσχουν και να, πιστέψουν ότι μπορούν να διαμορφώσουν και αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και ασκώντας τα πολιτικά τους δικαιώματα, αλλά και αντιμετωπίζοντας το δημοκρατικό έλλειμμα και τα υψηλά ποσοστά αποχής. Τον Αύγουστο του 2011 το Ευρωβαρόμετρο αποκάλυψε κάποια νούμερα και το Σεπτέμβριο του 2011 αποκάλυψε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ε, δεν ξέρουν πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες ποια είναι τα δικαιώματά τους. Στην Κύπρο, στη χώρα μου, ο κόσμος απάντησε ότι το 94% μάλιστα αυτών απάντησαν δεν ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει τον να μετακινούνται ελεύθερα και να ζουν ελεύθερα σε μια άλλη χώρα. Γιατί δικό στη χώρα μου ε, δεν υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση. Είναι μια έκθεση λοιπόν πολύ σημαντική, με πολλές προκλήσεις ε, για όλους μας αλλά και για τους Κύπριους, οι οποίοι θα αναλάβουν και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμεινο του 2012. Περιμένω λοιπόν να συνεργαστώ με τους κοιόδες εισηγητές, με την Κομισιόν, την Πολωνική Προεδρία και την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία, ούτω ώστε να προτείνουμε συγκεκριμένε δράσει. Βεβαίω, χρειαζόμαστε συνεργασία μεταξύ μα, τη βοήθεια όλων, αλλά όλα αυτά τα βήματα θα τα διανύσουμε πολύ προσεκτικά, θα διατυπώσουμε προτάσει με συγκεκριμένα μηνύματα, με συγκεκριμένο περιεχόμενο, για να υπάρξει αυτή η επικοδομητική συνεργασία. Περιμένω, την περιμένω και πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα η έκθεση για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδοπούλου. Υπάρχουν κάποια μέλη τα οποία θέλουν να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Σόμπορ καταρχήν. Προσπαθήσω να μιλήσω στα Ουγγρικά. Η πρόταση αυτή λοιπόν για το έτος των Ευρωπαίων πολιτών το 2013 δεν έχει σαν στόχο μονάχα να προωθήσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να διατυπώσει μια σειρά από σημαντικούς στόχους. Γνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε σχέση με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, σε σχέση με την πρόσβαση σε υγεία και άλλες υγειονομική περίθαλψη και άλλες ε, κοινωνικές υπηρεσίες πριν από ένα χρόνο ένα κράτος μέλος ένα κράτος μέλος εμπόδισε την ελεύθερη μετακίνηση του Προέδρου ενός άλλου κράτους μέλους. Δεν μπόρεσε ο Πρόεδρος ενός άλλου κράτους μέλους να μπει στο έδαφος του. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να πληροφορούμε συγχρόνω σε αυτού και αλλήλου και να υπάρχει μια πλήρη συζήτηση μεταξύ των πολιτών για την ελευθερία διακίνησης. Το κείμενο είναι θαυμάσιο, όπω είπε και ο πρόεδρο. Πρέπει να υπενθυμίσω όμω ότι όλα αυτά συνάπτονται και με το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη και τη στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πλευρά του ΕΛΚ και ως ο εισηγητής. Θέλω να πω ότι υποστηρίζουμε πλήρως την πρόταση της εισηγήτριας και ευχαριστούμε επίσης και την Κομισιόν. Και μετά πέθανε. Mr. Sober. Ευχαριστώ κύριε Σόμπορ, ναι. Μα. Κύριε Γκόντς. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την πρόταση αυτή. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχουμε μια εκδήλωση που θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να νιώθουν ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Αλλά θέλω να σας πεθυμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην δημιουργήσουμε περαιτέρω φρούδες, ελπίδες και απογοητεύσεις στο μέλλον με το να καθυστερήσουμε την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ζώνη του Σέγγεν. Αυτό είναι ένα κεφαλαίωδες θέμα ελεύθερης κυκλοφορίας και φέτος επίσης αντιμετωπίσαμε προβλήματα με την επανεισαγωγή των τελωνιακών ελέγχων σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι τα πράγματα που μαθαίνουν οι πολίτες μας κάθε μέρα γνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προσκόμματα για την ελεύθερη εγκατάσταση για να πάει σε άλλη χώρα, για να πάει κανείς να σπουδάσει σε μια άλλη χώρα, να πάει να εργαστεί κάπου αλλού. Μπορεί κανείς να πληροφορήσει τους πολίτες μας για τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά του και για το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προσκόμματα, τότε το έτος αυτό θα είναι πολύ επιτυχέ. Αλλιώ μπορεί να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη ματέωση και απογοήτευση. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος και δίνει το λόγο στην κυρία Λάντφορντ. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο θα μπορούσε να είναι κατά ενό τέτοιου έτου για τον Ευρωπαίο πολίτη. Δεν μου αρέσει να γκρινιάζω και να είμαι αρνητική, αλλά Έχω υπηρετήσει και σε αυτή την Επιτροπή και στην Επιτροπή των Αναφορών αρκετό καιρό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το σύνολο των προβλημάτων όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας στην διακίνηση. Τότε, αφού πετύχουμε την εφαρμογή της οδηγίας, θα πρέπει να γιορτάσουμε ένα τέτοιο έτος. Ξέρω ότι ακούγεται αυτό κάπως, μ, πώς να το πω, πώς να το πω έτσι πικρόχολο, αλλά θα κοστίσει χρήμα ο εορτασμός. Όμως, το θέμα είναι ότι υπάρχουν εδώ πέρα πραγματικές δυσκολίες για τα φυσικά πρόσωπα. Κάθε τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να Προσφύγεται την παραβάση και όλο και κάτι γίνεται. Εγώ θα ήθελα να γίνω ακόμα περισσότερα, αλλά ρίχτε μια ματιά στο τι προβλήματα μας λένε οι ψηφοφόροι σχετικά με την οδηγία του άρθρο 10 όσον αφορά τη μόνιμη παραμονή σε μια χώρα, τι γίνεται με τις ε, οικογένειες, με τους τις συζύγους, των, των, των, των μεταναστών ε, από τρίτες χώρες, τι γίνεται, τι γίνεται με τα ζεύγια ομοφιλοφίλων που προσπαθούν να έχουν την αμοιβή αναγνώριση όταν από μια χώρα πάνε σε άλλη και να έχουν αναγνωριστεί, χάνουν το προνομίο αυτό. Πάρα πολύ σημαντικά θέματα μπαίνουν τώρα εδώ πέρα. Κληρονομικού δικαίου, φορολογικού δικαίου κλπ. Πολλέ φορέ είναι και θέμα επιμέλεια και δαιμονία παιδιών και έχουμε τεράστια ζητήματα και μα είπε η Πολωνική Προεδρία ότι τα βλέπει όλα στρογγυλά και θα ήθελα να ξέρω εάν και η Πολωνία έχει εφαρμόσει με επιτυχία την οδηγία εκείνη του 4. Ίσως το έχει καταφέρει, δεν ξέρω. Ισχύει αυτό. Και για τα θέματα οικογενειακού δικαίου, λοιπόν, αν κάνουμε τέτοιο εορτασμό δίνουμε την εντύπωση ότι εορτάζουμε επιτυχία. Επιτυχία που όμως δεν έχει επιτευχθεί, δεν έχει γίνει. Τόσα χρόνια περάσαν, 7 χρόνια και πριν την οδηγία του 4 προηγήθηκε ένας όγκος νομολογίας, αποφάσεων που δεν πιάσαν τόπο. Δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση επομένως με την πλήρη έννοια της φράσης του όρου. Μου το λένε ψηφοφόροι μου. Άρα, ας κάνουμε κάτι πριν πάμε στον εορτασμό. Συγγνώμη για αυτή την κρίνια, αλλά νομίζω ότι είναι άστοχο του εορτασμό. Εκτό αν χρησιμοποιηθεί σαν ευκαιρία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι γίνεται για το, το πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Και έτσι να του ε, ενθαρρύνουμε να μας βομβαρδίσουν εμάς με αναφορές και την Κομισιόν με καταγγελίες. Συμπαθάτε με, αλλά έτσι έχει κατάσταση ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Βερζιάτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ, όπως και η κυρία Λάτφορντ και εγώ θα ήθελα να πω ότι με τον εορτασμό αυτού του έτους για τον πολίτη να μην περιοριστούμε στην ενημερωτική συμφωνία πάνω στην ε, είτε το ευρωπαϊκό πολίτη και στα προνόμια τα οποία αυτή συνεπάγεται διότι θεωρώ ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα του Ευρωπαίου πολίτη είναι το ότι αυτό παραμένει, διότι αυτή παραμένει ένα συμπλήρωμα της εθνικής ιδιότητας του πολίτη, της Ιθαγένειας. Αν κανείς δεν έχει την ηθαγένεια κράτους μέλους, τότε δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, θα πρέπει να τεθεί το εξής ερώτημα. Τι νόημα έχει να είναι κανείς Ευρωπαίος πολίτης. Εάν θέλουμε να ξαναποκτήσουν την εμπιστοσύνη του προ τα θεσμικά όργανα Ευρωπαίοι, τότε θεωρώ ότι αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ βασικό. Επίσης, υπάρχει θέμα ερμηνείας του όρου ιδιότητα του πολίτη. Άρα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι, εάν δεν υπάρχει, μία μελέτη του τι νόημα έχει ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη ει κάθε κράτο μέλο. Εγώ είμαι Γαλλίδα και στη Γαλλία αυτό είναι διαρκέ θέμα συζήτηση, όπω άλλωστε και άλλα πολιτικά θέματα. Αυτή η παλιά ιστορία τη Γαλλική Επανάσταση. Όμω θα πρέπει να προβληματιστούμε πραγματικά. Τι πάει να πει ε, αυτή η ιδιότητα. Συνήθως λέμε ότι δεν απονέμεται, αλλά αναγνωρίζεται η ηθαγένεια, η ιδιότητα του πολίτη. Οπότε πέραν αυτής της επίσημης και τυπικής αναγνώρισης που συνοδεύεται και από την ελευθερία της διακίνησης έχουμε και κάποια άλλα δικαιώματα και καλύτερη αναγνώριση της ελευθερίας έκφρασης που απορρέει. Οπότε με εκπλήσει το ότι στην ανακοίνωση αυτή και είναι να σας πω ακριβώς αυτό, αυτό το οποίο με ενόχλησε. Λέει ότι σε περίοδο κρίσης ε, είναι ε, ε, πολύ πιο σημαντική παρά ποτέ η ιδιότητα αυτή και θα πρέπει επομένως να υποστηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις και θα πρέπει με δυναμικό τρόπο να εμπλακούν οι Ευρωπαίοι πολίτες αυτές. Και νομίζω ότι ακριβώς με τέτοιο ορισμό της κοινότητας του Ευρωπαίου πολίτη δεν θα πάει μπροστά η υπόθεση αυτή. Και επίσης τώρα κατακλείδη ότι εκπλήσωμε μια που δεν συζητήθηκε η πρωτοβουλία για τη ιδιότητα του Ευρωπαϊκού Πολίτη, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι μια λεπτομέρεια που είναι πάρα πολύ σημαντική, ούτως ώστε να υπάρξει μια αυθεντική κατάσταση ηθαγένειας ευρωπαϊκής ιδιότητας πολίτη. Νομίζω ότι... Merci, Εντάξει, λέει ο Εγώ ως τελευταίος ομιλητής, λέει ο κ. Μπόντς, νομίζω ότι το κείμενο αυτό είναι πολύ καλό. Θα ήθελα να αναφέρω αυτά τα οποία είπε η κυρία Γκόντς και η Βαρονέσα τη της Στο παρελθόν έχουμε κάνει εκθέσεις για το ευρωπαϊκό έτος του Α, του Β, του Γ. Γενικά έχουν δημιουργήσει κάποιες υψηλές προσδοκίες και το αποτέλεσμα όμως είναι απογοητευτικό γιατί έχουμε σταθεί μονάχα σε γενικότητες. Νομίζω ότι Μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα για, για τους εξής λόγους. Υπάρχουν βέβαια γενικότητες, αλλά θα πρέπει να δοθούν και πληροφορίες για συγκεκριμένα δικαιώματα. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το παραμελεί στο Κοινοβούλιο. Είναι πολύ θετικό, είναι πολύ θετικό να προωθήσουν μια θετική αντιμετώπιση. Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου όμως θα πρέπει επίση να αντιμετωπίσουν και ουσιαστικά θέματα, τα θέματα όπου δεν ισχύει η ελεύθερη κυκλοφορία και δεν γίνονται σεβαστά τα πολιτικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μίλησε για τους νέους ε, ε, αποφύτους η κυρία Παπαδοπούλου που έχουν πρόβλημα να κινούνται μέσα στην Ευρώπη σε μια εποχή λιτότητας. Μπορούμε εδώ να αναφέρουμε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και γι' αυτό διαφωνώ με την κυρία Λάτφορντ για αυτά που είπε με το να αναφέρουν αυτά τα προβλήματα, <clears throat> δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Δεν μας στείλουν περισσότερες ε, επιστολές και email. Το... Οι πολίτες ξέρουν ποια είναι τα προβλήματα. Ξέρουμε ότι η λύση δεν μπορεί να δοθεί σε πολλά προβλήματα εδώ, παραδείγματος χάρη για την καθυστέρηση ένταξης Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Όλα αυτά μπορούν όμως να βοηθηθούν αν πάρουμε στα σοβαρά αυτή την έκθεση. Η ομάδα μας θέλει να πάρει αυτή την έκθεση στα σοβαρά και να τονίσει που βρισκόνται ακόμα συνεχιζόμενα εμπόδια για την <clears throat> ελεύθερη κυκλοφορία και την πρόσβαση. Κύριε Μπρόγκς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαρόσο αναφέρθηκε προηγουμένως ότι είχε πει ότι ο λόγος ύπαρξης της Ευρώπης είναι να δώσει την δυνατότητα στους πολίτες να έχουν συμμετοχή. Μάλλον να έχουν συμμετοχή οι ευρωκράτες είναι αυτό το οποίο γίνεται όλο και λιγότερο οι ευρωκράτες δεν ακούν την, την ε, άποψη των πολιτών. Όταν δεν τους αρέσουν αυτά που λένε οι πολίτες λένε ότι είναι λαϊκισμός αυτά που λένε και όχι δημοκρατία. Όταν θέλουμε να πληροφορήσουμε τους πολίτες αυτό το οποίο ελέγχθηκε πολλές, πολλές φορές σήμερα το απόγευμα, μιλάνε πάρα πολύ για συγκεντρωτική επικοινωνία. Όλα αυτά βασίζονται στην εντύπωση ότι η αντίσταση στο ευρωπαϊκό εγχείρημα προέρχεται από την έλλειψη πληροφόρηση και την άγνοια. Μπορείτε να το λέτε αυτό πληροφόρηση, για μένα είναι προπαγάνδα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πληρώνεται αυτή η προπαγάνδα από δημόσια κονδύλια. Η υπηκότητα είναι μια νομική σχέση μεταξύ ενός κράτους και των υπηκόων της. Εμείς ξέρουμε, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος. Αν υπάρχει μια υπηκότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα πρέπει να γίνει κράτος. Μα θέλουμε να καταστρέψουμε την ανεξαρτησία και την κυριαρχικότητα των κρατών μελών βήμα με βήμα με έναν τρόπο αδιόρατο. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και έχουμε και τη συνάντηση των συντονιστών αμέσως μετά. Σας κάνω έκκληση να μην το ξεχνάτε αυτό για να ολοκληρώσουμε τέλο πάντων αυτή τη συζήτηση. Ο κύριος Μούλτερ, πολύ σύντομα πρόεδρε. Κάθε λέξη που είπε η Κομισιόν και το Συμβούλιο με βρίσκει σύμφωνο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή συνεργασία και μέχρι τη μέρα που θα πεθάνω θα παραμείνω πεπισμένος Ευρωπαίος. Αλλά έχω μία αίσθηση ότι ξεχνάμε άλλα πράγματα που είναι σημαντικά στην Ευρώπη, την ε, απασχόληση, πολύ πιο σημαντικά. Και διαρωτώ με, τα προηγούμενα χρόνια τι καταφέραμε. Ούτως ή άλλως κάθε χρόνο είναι μια... έχουμε ένα ειδικό καθήκον, είναι μια ειδική χρονιά κάθε χρόνο. Και παρά τις προσπάθειες τα αποτελέσματα είναι μηδαμινά. Ε, ίσως κάνω λάθος, αλλά αυτή είναι η αίσθησή μου. Να δώσουμε ξανά τον λόγο στην Κομισιόν, η οποία ξεκίνησε με μια παρουσίαση, αλλά σας, σας παρακαλώ να αφήσετε και ένα λεπτό για τον Πολωνό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιαζίνσκι ούτω ώστε να απαντήσει κάποιες από τις ερωτήσεις που απευθύνονταν προς το Συμβούλιο. Θέλετε να πάρετε το λόγο κύριε Γιζίνσκι, ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να απαντήσω σε μια ερώτηση που έγινε προς το Συμβούλιο. Από όσο θυμάμαι, από τις πληροφορίες που λάβαμε από την Κομισιόν για αυτά τα θέματα μέχρι στιγμής, επιβεβαιώνεται ότι η χώρα που ασκεί σήμερα την Προεδρία στο Συμβούλιο δεν έκανε παράβαση αυτή της οδηγίας. Μιλάω για το πώς εφαρμόστηκε αυτή η οδηγία στη χώρα μου. Αλλά μπορώ να επανέλθω με περισσότερες πληροφορίες και να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για την πρακτική που ακολουθούμε και για την εφαρμοστέα νομοθεσία. λαμβάνω υπόψη μου όλα τα θέματα τα οποία προωθεί η Κομισιόν. Είμαι στη διάθεσή σας να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά σας απογοητεύω. Δεν υπάρχει διαδικασία που παραβάσει εναντίον μας για τα θέματα που αναφέρατε. Ευχαριστώ κύριε Γιζίνσκι που σέβεστε και το χρόνο. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος κι εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Για τους ευρωβουλευτές που εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την πρόταση της Κομισιόν. Θα ήθελα να απαντήσω συνολικά, σφαιρικά, στις ερωτήσεις που μου απευθύνθηκαν. Φυσικά, υπάρχουν τομείς όπου η άσκηση των δικαιωμάτων δεν είναι πλήρης. Αλλά ξέρουμε ότι είναι μια διαδικασία εν εξελίξει Και ο τελικός στόχος είναι να έχουμε δικαιώματα που τα ασκούμε πλήρως ελεύθερα απαντώ στην κυρία Λάτφορτ. Τους έξι τελευταίους μήνες, δέκα διαδικασίες επί παραβάση δρομολογήθηκαν σε σχέση με αυτά που προβλέπει η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία. Θέλω να απαντήσω στην κυρία Βερζιά, η οποία είπε ότι συνδέσαμε την κρίση με την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταξύ άλλων. Φυσικά, σε περίοδους κρίσης υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης. A gap of confidence, όπως λέμε και σε καλά γαλλικά, που υπάρχει μεταξύ των πολιτών και του πολιτικού επίπεδου, πρέπει να το καλύψουμε και ακριβώς η πρότασή μας αυτό έχει στόχο, να καλύψει αυτό το χάσμα σε ό,τι αφορά την ε, εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, την διαιώνισή τους. Υπάρχει μια μελέτη η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, η οποία σημαίνει άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών και κυρίως τι σημαίνει η ενεργή ηθαγένεια. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα είναι έτοιμα στο τέλος του 2011 και θα σας παρουσιάσουμε και μία έκθεση στην ε, Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτή την πρόταση πρέπει να, το δει, να τη δείτε ως καταλήτη. Η δράση μας δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον τομέα της επικοινωνίας. Υπάρχουν και άλλες διαστάσεις των δικαιωμάτων των πολιτών, φερρυπίν των δικαιωμάτων των πολιτών ως καταναλωτές, που θα πρέπει επίσης να μπορούν να ασκούνται στα πλαίσια αυτού του ευρωπαϊκού έτους των Ευρωπαίων πολιτών. η δράση μας δεν είναι προπαγάνδα. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Είναι και ενημέρωση και επικοινωνία. Επικοινωνία σημαίνει ε, και ενημέρωση προς τις δύο κατευθύνσεις. Υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο διαβιβάζεται προς τους πολίτες, αλλά ακούμε και όλα τους πολίτες τις απαντήσεις τους. Και η, επικοινωνία, η ανακοίνωσή μας αυτή, συγγνώμη, δεν ε, διαπνέεται από ένα πνεύμα λαϊκίστικο, από ένα πνεύμα προπαγάνδας, αντίθετα από αυτό που είπατε, αντίθετα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και θέλει να ενημερώσει τους πολίτες για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι απάντησα στις ανησυχίες και στα ερωτήματα με όσο τον πιο λακωνικό τρόπο. Ευχαριστώ. Η κυρία Παπαδοπούλου για την τελευταία παρουσίασή της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. αυτή η έκθεση μπορεί να παίξει το ρόλο του καταλήτη, ούτω ώστε να καταλάβουμε καλύτερα με ποιον συνομιλούμε. Σε αυτή την έκθεση πρέπει να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες δράσεις. Δεν θα πρέπει να έχουμε γενικολογίες, ούτε απλούς εορτασμούς με τις τροπολογίες μας. Θα πρέπει να, ασκήσουμε, να μιλήσουμε για το δικαίωμα Ελεύθερη κυκλοφορία παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορούμε να το εξασφαλίσουμε αυτό το δικαίωμα, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα εργασίας, ιδίως για τους νέους που αντιμετωπίζει το φάσμα της ανεργίας, πώς θα έχουμε καλή ποιότητα ζωής σε περίοδο κρίσης και πώς θα έχουμε ίσες ευκαιρίες για όλου, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει χάσμα ανάμεσα σε αυτού που ζουν στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης ή στις χώρες της Μεσογείου και του Νότου της Ευρώπης. Αυτό που θα συζητήσουμε λοιπόν είναι πώς θα συνεργαστούμε ούτω ώστε η ευρωπαϊκή ηθαγένεια να είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Τελειώνει εδώ πέρα η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Παρακαλώ όλους όσους είναι συντονιστές να παραμείνουν στην αίθουσα γιατί συνεχίζεται για αυτούς η συνεδρίαση. Οι υπόλοιποι να αποχωρήσουν. siamo un po' in ritardo. Perché? No. Eh? Eh? Credo di sì, che alle 6.30 dobbiamo finire.